Good afternoon, colleagues. Welcome to our meeting today. First of all, I have to address the agenda issue. Καλησπέρα συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στη σημερινή μας συνεδρίαση. Θα ήθελα καταρχάς ε, να συζητήσω να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεώρησε πω εγκρίνεται το σχέδιο μέσα διάταξη. Το πρώτο σημείο στην ημερησία διάταξη είναι μια ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο κ. Κατάινεν, Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς τον Αντιπρόεδρο κύριο Κατάινεν γιατί είναι πάντα διαθέσιμος να έρθει στην Επιτροπή μας και να συζητήσουμε πολύ σημαντικά θέματα και για την Επιτροπή μας αλλά και για την Κομισιόν. Η σημερινή ανταλλαγή απόψεων θα αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό και το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι μια πολιτική προτεραιότητα και για εμάς και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χωρίς λοιπόν καθυστέρηση θα δώσω αμέσως το λόγο στον Αντιπρόεδρο κύριο Κατάιναν και θα του θα... ζητήσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εξωτήμα μέλη σας. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε και πάλι να συζητήσουμε μαζί διάφορα ζητήματα. Αυτή τη φορά θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό και πιο συγκεκριμένα το ε, σχέδιο εργασιών. Στις 30 Νοεμβρίου περασμένου Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε λοιπόν το ε, πρόγραμμα εργασιών για την περίοδο 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό, ε, μαζί και με άλλα συναφή μέτρα. Αυτό αποτέλεσε τιμήμα ε, του ευρωπαϊκού πακέτου για τα οικολογικά ζητήματα που έχουμε διαμορφώσει για τους Ευρωπαίους πολίτες και σίγουρα σε αυτό το ευρύτερο πακέτο η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό ήταν ε, μία από τις πιο παρεξηγημένες ε, νομοθετικές προτάσεις που είχαμε κάνει, γιατί πολλοί μας έχουν ε, επικρίνει και έχουν επικρίνει αυτή την οδηγία, γιατί λένε ότι επικεντρώνεται σε πολύ μικρά και δευτερεύοντα ζητήματα χωρίς ε, να ε, δίνει έμφαση, την απαραίτητη έμφαση στα μεγάλα και σημαντικά. Ενώ στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο. Γι' αυτό και θεωρώ ότι έπρεπε να εντάξουμε το πρόγραμμα ΣΥΟΝ για τον οικολογικό σχεδιασμό στο ευρύτερο πλαίσιο, γιατί νομίζω ότι αυτό ενισχύει ε, και τονίζει τη σημασία του οικολογικού σχεδιασμού και της οικολογικής επισήμανσης. Γιατί όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την καταπολέμηση της κλιματική αλλαγή, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ως ε, τμήμα τη ευρύτερη στρατηγική μας. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε και το θέμα τόσο καλά που δεν χρειάζεται και εγώ να σας εξηγήσω ε, τα βασικά. Όπως ξέρετε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την οπτική γωνία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων για να δούμε τι ευκαιρίες ε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε για αυτά τα δύο μέτρα. Ε, για την εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν και να είναι καλά ενημερωμένοι για να μπορούν να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικά αυτά τα μέτρα για την οικολογική επισήμανση. Ε, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών, BEUC, αναφέρει ότι η μέση εξοικονόμηση ενέργειας ε, κάθε νοικοκυριού θα είναι περίπου 450 ευρώ. Η Επιτροπή υπολογίζει ότι θα είναι 500 ευρώ η εξοικονόμηση ε, λόγω της και χάρη στην οδηγία αυτή, αλλά βρισκόμαστε περίπου στο ίδιο μήκος Όταν λοιπόν οι καταναλωτές ε, θα είναι πιο ενημερωμένοι, και θα μπορούν έτσι να επιλέγουν ε, τέτοια πιο οικολογικά προϊόντα, θα έχουν και την αντίστοιχη ε, οικονομική εξοικονόμηση. Η οδηγία δίνει τις ευκαιρίες όμως και στον κλάδο των επιχειρήσεων, γιατί αξιοποιώντας τον οικολογικό σχεδιασμό και την οικολογική επισήμανση, δημιουργούμε ταυτόχρονα και μία ενιαία αγορά όπου όλα τα προϊόντα είτε έχουν κατασκευαστεί στην Ευρώπη είτε σε τρίτες χώρες θα πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια. Η ανατροφοδότηση που έχουμε λάβει από τον ιδιωτικό κλάδο, από τους κατασκευαστές δηλαδή, είναι πολύ ενθαρρυντική, γιατί και αυτοί που τα κατασκευάζουν ε, ε, εποφελούνται, αλλά και αυτοί που είναι καταναλωτές τέτοιων προϊόντων. Και έτσι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τα. Και ακούμε πολύ πιο ενθαρρυντικά σχόλια και από την πλευρά της ε, βιομηχανίας σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια. Ο οικολογικός σχεδιασμός έχει ε, τεθεί σε ισχύ εδώ και 11 χρόνια. Έχουμε περίπου 30 ε, υποχρεωτικούς κανονισμούς ε, που ορίζουν ελάχιστα όρια ενεργειακής απόδοσης ή μέγιστον επιπέδων θορύβου, χρήσης ύδατος κτλ. Περίπου 15 από αυτές τις κατηγορίες προϊόντων. Επίσης, ε, υπόκειται στον υποχρεωτικό, στην υποχρεωτική ενεργειακή επισήμανση, στη γνωστή πυραμίδα A G. με τη χρήση αυτών των 30 ε, κατηγοριών προϊόντων γίνεται ήδη εξοικονόμηση ενέργειας ίση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας στην Ιταλία. Κάθε χρόνο λοιπόν, όχι μια φορά τώρα, κάθε χρόνο η ενεργειακή μας ε, εξοικονόμηση ισούται με την ενεργειακή κατανάλωση της Ιταλίας. Μόνο και μόνο χάρη στα μέτρα του οικολογικού σχεδιασμού. Για να τα αναφέρουμε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, αυτό ισούται με 1,3 δις βαρέλια πετρελαίου. ή 130 πυρηνικά εργοστάσια. Είναι λοιπόν τεράστια τα ωφέλη. Είπα λοιπόν και στην αρχή ότι μας επικρίνουν ότι η οδηγία οικολογικού σχεδιασμού είναι ίσονος ε, σημασίας ε, γιατί δεν επηρεάζει ε, το μεγάλο διακύβευμα, αλλά αυτό δεν ισχύει, βλέπετε. Μπορεί κάποιος να νομίζει ότι ο, ο, βραστήρας και ο στεγνοτήρας χεριών δεν έχει μεγάλο αντίκτυπο, αλλά αν το δούμε συνολικά και τη συνολική εξοικονόμηση ενέργειας, τότε είναι πραγματικά πολύ σημαντικές οι συνέπειες η νέα, μάλλον το νέο πρόγραμμα εργασιών για την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού που υιοθετήθηκε στα τέλη της περασμένης χρονιάς προσέθεσε 7 στοιχεία στον κατάλογο του οικολογικού σχεδιασμού συστήματα αυτοματισμού στην κατασκευή, ηλεκτρικοί βραστήρε, ενελκυστήρε, τεχνοτήρε χεριών, ηλιακοί συλλέκτε, inverters και εργαλεία καθαρισμού υψηλή πίεση μεταξύ άλλων. Όταν τα έχουμε υλοποιήσει όλα αυτά και αυτά τα προϊόντα έχουν μπει στον κατάλογο κανονικά, ε, θα έχουμε ξεκονώσει με ενέργειας αντίστοιχη με την κατανάλωση ενέργειας της Σουηδίας σορευτικά πέραν της Ιταλίας. ...50.000 λιγότερες ανεμογεννήτριες ή 30.000 λιγότερα πυρηνικά εργοστάσια ή 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου λιγότερο για την Ευρώπη. Τεράστια λοιπόν η σημασία της οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού. Από εδώ και στο εξή. Ε, η ε, θεωρία της κυκλικής οικονομίας ε, για την επανάχρηση και επαναξιοποίηση θα μας απασχολήσει πιο συγκεκριμένα για να θέσουμε σε εφαρμογή τους στόχους για την κυκλική οικονομία. Κύριε Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ. Αυτό που ήθελα να πω εδώ είναι ότι αυτές οι δύο νομοθετικές προτάσεις ε, είναι ιδιαίτερα υποφελείς, αλλά μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο αν εισαγάγουμε και τις αρχές της επανάχρησης ε, και επαναξιοποίησης και ε, καλύτερης των προϊόντων και αν τα ενσωματώσουμε όλα αυτά στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο πρέπει, καλά τα συζητάμε μεταξύ μας, αλλά πρέπει να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και των πολιτών, γιατί όλοι θέλουν να ακούσουν ε, τα στοιχεία, τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα ε, μέσα αυτών των ε, μέτρων που είναι αξιοθαύμαστα και αυτό δείχνει ε, πόσο ωφέλιμο είναι αυτό το πλαίσιο. γιατί μόνο η ολοκληρωμένη Ευρώπη ε, μπορεί να τα πετύχει όλα αυτά. Όταν είμαστε κατακαιρματισμένοι δεν μπορούμε να έχουμε αυτές, αυτή την εξοικονόμηση και αυτές τις ευκαιρίες. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Να σχολιάσω κι εγώ λέγοντας ότι προφανώς πρόκειται για ένα από τα στοιχεία που η Ενωμένη Ευρώπη φέρει προς τα θέμενη αξία και είναι ζητήματα που απασχολούν και την Επιτροπή μας. Γι' αυτό ήταν και πολύ επίκαιρη η παρατήρηση που κάνατε προηγουμένως. Είναι σημαντικό. Σα ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την παρουσίασή σας. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στου συναδέλφου. Ο κύριος Λίζα πρώτος. Ο κύριος Πέτερλε πρέπει να φύγει νωρίς, γι' αυτό λοιπόν θα του δώσω το λόγο και μετά θα μιλήσω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, για να μην είμαστε τόσο γραφειοκρατικοί, την άλλη φορά δεν θα χρησιμοποιήσω κατάλογο. Κύριε Πέτερλε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω τα εξή. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα συνεχίσω στη μητρική μου. Οπότε βάλτε τα ακουστικά σας. Το είναι το καλύτερο μέρος ε, της σημερινής ε, ημέρας. Ακούμε ε, για κάτι το οποίο λειτουργεί καλά. Χαίρομαι που βλέπω ότι ε, λειτουργεί αυτό το ευρύτερο πλαίσιο και το στηρίζω. Είναι η καλή προσέγγιση που έχετε. Πρέπει λοιπόν ε, να δούμε τον ε, πλήρη ε, κύκλο ζωής των προϊόντων αυτών. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα σημαντικό τμήμα του πράσινου πακέτου. Όπως έχω πει, ο καταναλωτής μπορεί να το κατανοήσει, μπορεί να το αξιολογήσει, να δει αν λειτουργεί ή όχι. Σας εύχομαι Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια της εργασίας σας. Ε, βλέπω ότι έχετε τη σωστή προσέγγιση και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Πώς ε, βλέπουν οι συνάδελφοί σας ε, το ρυθμιστικό πλαίσιο. Όταν μιλούμε για νέα καινοτόμα στοιχεία από αυτά, συνήθως εξετάζουμε το κόστος, το κόστος του νέου ρυθμιστικού πλαισίου και θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η γνώμη των συναδέλφων σας. Πώς θα ε, προωθήσετε αυτό το project και νομίζω πρέπει να το χειριστείτε σωστά. Ευχαριστώ κυρία Ντάλη. ευχαριστώ. Ix tajjeb niċċaraw u nenfasizzaw li l-Ewropa mhijiex l-uniku reġjun laqas li qiegħed jiffoka u jimbotta u jipromovi. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρώπη πραγματικά είναι ε, ο μοναδικός τρόπος να προαγάγουμε αυτή την έννοια της κυκλικής οικονομίας. Και όταν το εξετάζουμε βλέπουμε πολύ συχνά για παράδειγμα, ότι την Κίνα και ότι και εκεί υπάρχουν πολλά μέτρα και, μπορούν, και προσπαθούν να ε, προωθήσουν την κυκλική οικονομία και στην Κίνα δίνουμε μεγάλη έμφαση και στην ε, βιωσιμότητα και τον ε, κύκλο ζωής των προϊόντων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίως αν λάβει κανείς την υπόψη τη θέση της Κίνας σε ό,τι αφορά το Key Manufacturing Hub και στις ΗΠΑ ε, υπάρχει, ε, υπήρξε και μια συνδιάσκεψη για αυτό το ζήτημα και αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να συνεχίσει και η Ινδία σε αυτή την οδό της ε, κυκλική οικονομία, Αυτό θα είχε πάρα πολλά ωφέλη. 600 δις δολάρια θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν με αυτόν τον τρόπο. Και Εάν συνεχίσουμε να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην κυκλική οικονομία, έτσι μπορούμε να εξαλείψουμε και άλλους αρνητικούς ε, κλάδους, όπως είναι ε, η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Ε, αλλά να μειώσουμε και την ρήπανση και αυτό θα ωφελήσει γενικά και την δημόσια υγεία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού. Δύο ερωτήματα λοιπόν προς τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να μας δώσετε πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, θα υιοθετηθούν για να προσαρμόσουν ακόμη περισσότερο τις προποθέσει τη οδηγία στην κυκλική οικονομία. Και δεύτερον, πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με τι ΗΠΑ ό,τι αφορά την εποπτεία τη αγορά. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βελτιώσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κερκράντη. Να πεθυμίσω τα δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε ευχαριστώ που ήρθατε. Αυτά που είπατε για την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών είναι πολύ σημαντικά. Επιπλέον όμως πρέπει να ισχύσει αυτό και για τους υψηλόβαθμους πολιτικούς μας. Ο κ. το 2014 στην εκλογική εκστρατεία για την Ευρωβουλή έγινε αντικείμενο χλεβασμού για την ηλεκτρική σκούπα στην Ολλανδία. Και από τότε βέβαια έχουν περάσει χρόνια και καταλάβαμε τέλος πάντων τι σημαίνει οικοσχεδιασμός, εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν θα πάω από τα στοιχεία που αναφέρατε, αλλά βλέπουμε ακριβώς το πόσο εύκολα αυτή η πολιτική μπορεί να γελιοποιηθεί και πόσο εύκολα μπορεί να πιστεί ο κόσμος αν δει το θέμα σοβαρά και καταλάβει τις τεράστιες ευκαιρίες που βρίσκονται εδώ. Και αυτό που έγινε με τον κύριο Τίμερμαν θα πρέπει να γίνει και με του αρχηγού κυβερνήσεων και εντό τη Κομισιόν και να αφορά και τον πρόεδρό τη. γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα. Δεν σημειώνουμε επαρκή πρόοδο, δηλαδή κολλάμε σε μια τεχνοκρατική διαδικασία και διαβάζω εδώ το σημείο 9, τη σελίδα 9 του εγγράφου με διάφορα τετραγωνάκια. Εντάξει, ξέρω δύο πράγματα για αυτό το θέμα, αλλά εδώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πολυλογία μόνο βλέπω και δεν βλέπω να πηγαίνουμε στο ψητό. Και από ό,τι κατάλαβα, βλέποντας και άλλα σχέδια, ας πούμε, οι προτάσεις για εφαρμογή αυτού του κανονισμού σε σχέση με τις οθόνες και και τις τηλεοράσεις είναι έτοιμη η νομοθεσία, αλλά υπάρχει συζήτηση εσωτερική στου βιομηχανίε για το τι πρέπει να κάνουμε. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε λοιπόν που βρισκόμαστε, πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά και να τολμήσουμε πολιτικά, γιατί δεν έχουμε την πολιτική πεποίθηση και την δύναμη να το κάνουμε αυτό. Οπότε αυτό είναι το κυρίω μου ερώτημα. Πότε, πότε λέω, πότε τέλο πάντων όλα αυτά θα γίνουν στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο, πέραν δηλαδή αυτή του τεχνοκρατικά απλά ρήματος. Ευχαριστώ. Επόμενος ο κύριε Άβαν. Ευχαριστώ που ήρθατε. Η Κομισιόν νομίζω έχει δείξει κάποια δυναμία εδώ σε αυτό το ζήτημα. Και αυτό αφορά και τη δικιά σας πολιτική οικογένεια, ο Τίμερμαν, ο Γιούνκερ κτλ πώς γελικοποιήθηκαν στις εκλογικές εκστρατείες. Σε αντίθεση με εμά που γνωρίζαμε την οδηγία, την ξέραμε και μπορούσαμε να πείσουμε τον κόσμο ότι είναι ήταν καλή οδηγία. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερη δέσμευση ώστε να περάσουμε επιτέλους στα αφαρμοστικά μέτρα, γιατί πραγματικά η οδηγία είναι πολύ καλή το ιδεολογικό της υπόβαθρο είναι πολύ καλό. Ο οικοσχεδιασμός λοιπόν είναι πολύ χρήσιμος για τους καταναλωτές. Να ξέρουν τέλο πάντων οι καταναλωτέ τι γίνεται με κατανάλωση ενέργεια, νερού, στα μπάνια, στα λουτρά. Και αυτά τα θέματα λοιπόν μας ανησυχούν και βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί ας πούμε τον οικοσχεδιασμό ας πούμε στα έξυπνα τηλέφωνα όπου εκεί πρέπει να έχουμε τον κατάλληλο σχεδιασμό, να έχουν την κατάλληλη μορφή, αυτά κλπ. κλπ. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τη χρήση των πόρων, ανθρώπινων πόρων, υλικών πόρων και τη χρήση του ώστε εδώ να κάνουμε κάτι το χρήσιμο. Θα μπορέσετε λοιπόν να μας διαβεβαιώσετε ότι επιτέλους θα γίνει κάτι και θα υποβάλλετε επιτέλους ένα σχέδιο το οποίο θα αποδεικνύει ότι τέλος πάντων ότι υπάρχει και βούληση, ότι υπάρχουν οι και ότι θα προχωρήσουν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντορνάνα. Ντορνάνο. Ντορνάνο, λέει πρόεδρος, διορθώνει. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αυτή η παρουσίαση του προγράμματος της Κομισιόν γίνεται ενώ συζητάμε αυτή την προγραμματισμένη αχρηστία των συσκευών. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με τη χρήση της ενέργειας, με την επισήμανση, με τις δυνατότητε που περιλαμβάνουν οι συμβάσεις κτλ. Όμως όλα αυτά ως πρωτοβουλίες αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και είναι δύσκολο να καθορίσουμε κριτήρια βιωσιμότητας και ενεργειακής κατανάλωσης αξιόπιστα. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά λοιπόν στα ανάντι, γιατί η μαζική παραγωγή αγαθών με χαμηλό κόστος αποτελεί την πηγή της χαμηλής τους βιωσιμότητας στη διάρκεια ζωής. Και η Κομισιόν ρωτώ θα υποστηρίξει μέτρα που θα παροτρύνουν τη χρήση προς τη σωστή κατεύθυνση ανταποκρινόμενη και σε κάποια κριτήρια ποιότητας. Και πώς έχετε εσείς αντιμετωπίσει ακριβώς το θέμα αυτό της βιωσιμότητας του κύκλου ζωής των προϊόντων σε σχέση με κάποιες χώρες οι οποίες είναι μεγάλη παραγωγή αυτών των προϊόντων. Χρειαζόμαστε λοιπόν προγράμματα αντικατάστασης αυτών των ελάχιστα οικολογικών προϊόντων με άλλα προϊόντα πιο οικολογικά, πέρα δηλαδή από την καταπολέμηση της κατάχρησης αυτών των προϊόντων. Σήμερα, ας πούμε, οι λάμπες ε, LED που θεωρούνται βλαβερές για την υγεία. Ε, θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται και με αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επίτροπε. Μήπως θέλετε να απαντήσετε στο πρώτο γύρο απαντήσεων. Ναι, και ρωτήσαν. Ευχαριστώ, λέει ο Επίτροπος. Να σας δώσω κάποια γεγονότα, μάλλον ενδιαφέροντα. Κάποια στοιχεία μάλλον. Αν δούμε την εξοικονόμηση ενέργειας που λέγαμε προηγουμένως για την Ιταλία ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της οδηγίας Είπαμε πριν ότι έχουμε εξοικονομήσει ίση με την ε, κατανάλωση στην ετήσια ενέργεια τη Ιταλία. Εδώ θα έχουμε λοιπόν και μια εξοικονόμηση 340 εκατομμύριων τόνων διοξιδίου άνθρακα. Λόγω και μόνο του οικοσχεδιασμού, του σχεδιασμού αυτών των προϊόντων, του οικολογικού. Μπορούμε να πετύχουμε λοιπόν μια μείωση εκπομπών διοξιδίου, άθρακα τεράστια. Χωρίς αυτήν την οδηγία λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τους καταναλωτές με τη δουλειά που γίνεται για το περιβάλλον. Θα έπρεπε να πιέσουμε για τη σωστή παραγωγή αυτών των προϊόντων. Και πρέπει να δούμε τώρα βεβαίως τι μπορούν να συμβάλλουν και τι μπορούν να κάνουν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, οι ίδιοι οι πελάτες αυτών των προϊόντων για να έχουμε σωστά αποτελέσματα. Ο κ. ρώτησε το πώς προσεγγίζουν την οδηγία αυτή οι υπόλοιποι συναδέλφοι μου. Κοιτάξτε, υπάρχουν αποκλείωσες τέλος πάντων προσεγγίσεις διαφορετικές. Η οδηγία αυτή νομίζω κερδίζει έδαφος και μετά από μια εντελεχή διαδικασία στην Κομισιόν βλέπουμε ότι έχει μια ισχυρή πολιτική στήριξη, μεγαλύτερη από ποτέ. Ίσως αυτή η εργασία, έστω και αν χρειάστηκε περισσότερο χρόνο, νομίζω ότι αποτελεί μια καλή πολιτική δουλειά με την κατάλληλη στήριξη. Είναι επίσης σημαντικό από αυτή την μακροσκελή διαδικασία Να πούμε ότι για πρώτη φορά υπάρχει τόσο ισχυρή τέλο στήριξη εκ μέρου τη Κομισιόν ώστε να προωθήσουμε ακριβώ τον οικοσχεδιασμό. Νομίζω ότι βέβαια όλοι εντάξει μπορούμε να πετύχουμε και περισσότερα όταν μιλάμε με τους πολίτες για αυτή την οδηγία και τα αποτελέσματά της. Ε, εμείς βέβαια δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα παραβιάζει θέματα η δικασία ανταγωνισμού, η δικαιώματα πολιτών κτλ. Εμείς θέλουμε απλά και μόνο τα προϊόντα τα οποία παράγονται να είναι ισοδύναμα, να δίνουν τη δυνατότητα λέει στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά τα προϊόντα αυτά και βεβαίως και η ίδια η βιομηχανία να έχει και αυτή έτσι μια ισοτιμία στον τομέα αυτό. Τώρα για το μέλλον της οδηγίας του οικοσχεδιασμού. Όπως είπα στην εισαγωγή μου, θέλουμε να αναπτύξουμε περισσότερο αυτό το εργαλείο. Δεν είναι απλό αυτό, έτσι. Όταν εντάσσουμε στοιχεία όπως κατά πόσο μπορεί κανείς να επισκευάσει ένα αντικείμενο ή η επαναχρησιμοποίησή του κτλ. κτλ. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε αναπροϊόν. Αλλά πάντως χαίρομαι γι' αυτό, γιατί φανταστείτε αν τα μελλοντικά κινητά τηλέφωνα θα ήταν πιο εύκολο να επισκευαστούν. Τότε ο καταναλωτής βεβαίως θα το αναβάθμιζε αντί να το πέταγε και να αγοράζει ένα καινούριο. Αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την απόδοση των πόρων. Εφ' λοιπόν, δεν θα κοιτάμε τα προϊόντα μόνο από τη σκοπιά της ενεργειακής απόδοσης, αλλά και από τη σκοπιά του κατά πόσο θα μπορούσε κανείς να εντάξει εδώ άλλες διαστάσεις στον κανονισμό πέρα δηλαδή της ενεργειακής απόδοσης. Στην οδηγία, συγγνώμη. Είμαι πάντως πεπισμένος ότι θα υπάρξουν αρκετά προϊόντα πάνω στα οποία θα μπορούσαμε να βάλουμε στόχους τέλο πάντων επαχρησιμοποίησης ή λειτουργικότητας κτλ. Αλλά αυτό δεν θα ισχύσει βέβαια για όλα τα προϊόντα ή με όλα τα προϊόντα. Επίσης, για την ευαισθητοποίηση στο υψηλότερο να το πολιτικό επίπεδο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Ότι δηλαδή αυτή η νομοθεσία ήταν αντικείμενο κατάχρησης για πολλά χρόνια και θέλωσε τα νερά αυτό. Οπότε δεν χρειάστηκε μόνο να πρασπιστούμε την, ε, το καλό όνομα του οικοσχεδιασμού, αλλά και να δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Και όπως είπα πριν, αυτό είναι από τα πιο ευκολονόητα θέματα, γιατί ακριβώς καταδεικνύει την σημαντική αξία της ευρωπαϊκής προσέγγισης και εγχειρήματο. Τέλος, τα κίνητρα. Τι κίνητρα θα μπορούσε να δώσει η Κομισιόν, να δημιουργήσει η ίδια η Κομισιόν για καλύτερη κατανάλωση. Νομίζω ότι ο ρόλος μας είναι να διασφαλίσουμε το ότι οι καταναλωτές θα λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όταν έχουν να κάνουν ή έχουν να λάβουν μάλλον αποφάσεις που αφορούν την κατανάλωση κάποιων προϊόντων. Η πληροφορία λοιπόν είναι ένα εργαλείο, η πληροφόρηση και επίσης μπορούμε να θεσπίσουμε και περιγραφές ποιότητας στα πλαίσια της οδηγίας για τον οικοσχεδιασμό. Τώρα, αλλά κίνητρα δεν βλέπω προ το παρόν. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος για το σχέδιο δράσης. Για φέτος σχεδιάζουμε αυτή την στρατηγική για τα πλαστικά. Επίσης θέλουμε να υπάρχει μια χρηματοοικονομική πλατφόρμα και άλλες συγκεκριμένε προτάσεις οι οποίες ε, προέρχονται από τον κλάδο. Οπότε προχωρά το σχέδιο δράσης και νομίζω θα οδηγήσει τελικά σε συγκεκριμένες προτάσεις. Όπως είπαμε και πέρσι στην προηγούμενη εμφάνισή μου εδώ, το σχέδιο δράσης βρίσκεται στις απαρχές του. Οπότε οι ευκαιρίες είναι τεράστιες εδώ σε αυτούς τους τομείς. Και βεβαίως εμείς έχουμε κάθε διάθεση να αποφεληθούμε από κάθε δυνατή ευκαιρία. Θα έχουμε και μέσα στη χρονιά και άλλες προτάσεις που αφορούν τα χημικά προϊόντα. Θα έχουμε νομοθεσία για τα απορρίμματα και για την κυκλική οικονομία θα έχουμε επίσης και ένα πλαίσιο εποπτείας Αυτά είναι τα, τα στοιχεία τα οποία θα μας απασχολήσουν φέτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από ό,τι βλέπω υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο. Υπάρχει κάποιος άλλος πέρα από αυτούς που το ζήτησαν. Ναι, ναι, συγγνώμη που δεν λάβατε το λόγο πριν, αλλά θα σας τον δώσω σε λίγο. Σας ευχαριστώ. Εκτός λοιπόν από την κυρία Ρίτ, υπάρχει κάποιος άλλος, ο κύριος Λίζα, ναι βεβαίως είστε στον κατάλογο. Κάποιος άλλος και εσείς. Μάλιστα, κλείνω ο κατάλογος των ομιλητών. Η κυρία Ριντ θα λάβει το λόγο ως συντονίστρια. Ξεχάσετε όμως να σηκώσετε το χέρι σας πιο πριν. Έχω μια ερώτηση για τον κύριο Πίτροπο. Θα με ενδιαφέρει πολύ ε, να μάθω περισσότερα για αυτό που είπατε, ότι κάθε χρόνο δηλαδή η ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη μειώνεται. Ε, γνωρίζετε κατά πόσο αυτό οφείλεται στην ε, βαριά βιομηχανία, κατά πόσο συνεισφέρει η διαρροή διεξιδίου άνθρακα. Τι γίνεται με τη βιομηχανία που πηγαίνει στην Κίνα και την Ινδία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ελίζα, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς κύριε Αντιπρόεδρε που ήρθατε εδώ, ευχαριστώ πολύ για την προθυμία που δείχνετε να έρχεστε πάντα και να μιλάμε. Οικολογικός σχεδιασμός λοιπόν, πριν από λίγο καιρό ενημερωθήκαμε για το πρόγραμμα, θα ήθελα να πω και εγώ λοιπόν, όπως είπε και η κυρία Ρίντο, ότι αυτό ακριβώ το μέσο θα εφαρμοστεί ε, ανεξαρτήτως ε, χώρος προέλευσης σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά, δηλαδή είτε σε εταιρείε από την Κίνα είτε από την Ινδία. Και εδώ έχουμε το πρόβλημα της διαρροής διοξιδίου του άνθρακα που ανέφερε και η κυρία Ριντ και είναι κάτι πάνω στο οποίο μας έχει ασκηθεί πάρα πολύ ε, κριτική. Τώρα, ορισμένα προϊόντα όπως οι τοθιέρες, οι φρυγανιέρες, τα κεφάλια του ε, ντους, οι, τους γέρες, αυτά εξαιρούνται και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί πρέπει με, να εξηγήσουμε στον καταναλωτή πώς ε, μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια, ότι πρέπει να εξοικονομήσει ενέργεια, αλλά δεν μπορούμε να περιορίζουμε κάθε του κίνηση. Τώρα δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται με ορισμένα ε, προϊόντα. Πώς θα καταφέρουμε δηλαδή να εφησυχάσουμε τους καταναλωτές, να καθησυχάσουμε τους φόβους τους για το ότι θα περιοριστεί, ε, θα περιοριστεί η ζωή τους με αυτές τις ε, νέες συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Σαλτεμόζο, ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας. Χαίρομαι πολύ που είστε ανοιχτό ε, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς την ανταλλαγή απόψεων. Η Επιτροπή μας ασχολείται εδώ και πάρα πολύ καιρό με μια έκθεση που ε, αφορά το να χρησιμοποιούμε περισσότερο διάφορα, διάφορες ηλεκτρικές συσκευές. Μας είπατε ότι θα Κοιτάξτε τα κριτήρια βιωσιμότητας κατά τομέα και ιδιαίτερα συγκεκριμένους τομείς. Όμως ε, σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα αναφέρεται επίσης ότι υπάρχει και για ορισμένα προϊόντα ένας χρόνος ζωής τρία χρόνια ή χίλιες ώρες, για παράδειγμα για τους λαπτήρες. Ο καταναλωτής πώς θα ε, μπορεί να γνωρίζει το χρόνο ζωής ενός προϊόντος πριν το αγοράσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλόρεντς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε, κύριε την Πρόεδρε. Ήδη έχουν γίνει πολλές καλές ερωτήσεις, ε, αλλά επιτρέψτε μου να επανέλθω στο αγαπημένο μου θέμα, την κυκλική οικονομία. Εξεπλάγει όταν είδα ότι θα χωρίσουμε τον κανονισμό REACH από την ε, στρατηγική διαχείριση αποβλήτων. Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Διότι η διαχείριση απορριμμάτων γενικότερα νομίζω πως συνδέεται απόλυτα με τους στόχους ε, του κανονισμού REACH. Δεν βλέπω όμως εδώ κάποια στρατηγική, κάποια περισσότερη ενημέρωση. Θα μπορούσατε να μας πείτε λοιπόν κάτι παραπάνω γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιούσο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίτροπε, μιλώ και μέρου του κύριου που, ο οποίος απουσιάζει λόγω πτήση. Ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε σήμερα εδώ, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, για να μιλήσουμε για τον οικοσχεδιασμό που έχει ένα ρόλο όσον αφορά την αλλαγή του Παραδείγματο στην Ευρώπη σε σχέση με την κυκλική οικονομία. Αποτελεί όμως και ένα στοιχείο κλειδί, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της Κομισιόν, για την εξοικονόμηση περίπου 500 ευρώ ανά νοικοκυριό ετησίως. Είναι χρήσιμο λοιπόν το στοιχείο στην εξοικονόμηση ενέργειας, στον περισμό των ρήπων, στην καταπολέμηση των παραγόντων που υποβαθμίσουν το κλίμα να σας ρωτήσω για τα ηλεκτρικά οχήματα. Προβλέπετε κάποιο, κάποια χρηματοδότηση ώστε να καταπολεμήσουμε την ρήπαση στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Επίσης προβλέπετε κάποιο σχέδιο οικονομικής στήριξης στους καταναλωτές ώστε να αντικαταστήσουν τα παλιά τους προϊόντα που ρηπαίνουν με νέα προϊόντα πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Κυρία Περτικάινεν. Ευχαριστώ πολύ. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό έχει ε, κάποιο πρόβλημα image αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν νομίζω πως ε, πρέπει να ρίχνουμε το φταίξιμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν ευθύνη και οι πολιτικοί σε, ε, στις... Ε, χώρες, τα κράτη-μέλη, αλλά και εμείς εδώ οι ευρωβουλευτές. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε πρώτα στον καθρέφτη πριν κατηγορήσουμε άλλους και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Θα ήθελα εγώ να σας ευχαριστήσω για τη δραστηριότητα που έχετε επιδείξει ε, σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες αναπάντητες ερωτήσεις για το μέλλον. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να δούμε κάποια μεγάλη αλλαγή ε, σε ό,τι αφορά την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού. Κάποια οριζόντια αλλαγή για ορισμένα αγαθά και στην ενία αγορά και αλλού. Είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε και με τα μη βιώσιμα εισαγόμενα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό τι δηλαδή συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς σκέφτεστε ε, να ενεργήσετε. Και μετά, ας αναφερθήκατε σε κάποιους δείκτες, σε κάποια πλατφόρμα ελέγχου, υπάρχει κάποιο σχέδιο που ξεπερνά την ε, απλή καθοδήγηση. Θα υπάρχουν δηλαδή κάποια δεσμευτικά κριτήρια δεδομένων των ε, προβλημάτων που όλοι γνωρίζουμε πως υπάρχουν εδώ. Και τέλος, θα μπορούσατε να μας πείτε ε, δύο λόγια για το πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το ΕΦΣΥ για εδώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χιάνς Καρσία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κομισιόν, με χαρά σας ξαναβλέπω για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως ο ανταγωνισμός. Θα θυμάστε την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε για την βελτίωση του, της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα. Σας είχα μιλήσει τότε για το food defense. Να επιμείνω λοιπόν σε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να στηρίξουμε ένα επιχειρηματικό κλάδο που μπορεί να δημιουργήσει θέσει εργασία και που βεβαίω είναι ανοιχτό σε συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη. Πρέπει όμως να παρέχει και κυρίως ασφάλεια στον καταναλωτή. Έχουμε αυτή τη στιγμή διάφορες ε, επιθέσεις, τρομοκρατικές κτλ. Τι καλύτερο λοιπόν μπορούμε να κάνουμε από το να ενισχύσουμε το food defense. Για το, λοιπόν, το άνοιγμα των αγορών, την απασχόληση κτλ. Τι καλύτερο από το να υποστηρίξουμε τη μηχανία αυτή με το food defense με τρόπο ώστε να αναγνωρίζεται από χώρε όπω η Ιαπωνία, η ΕΕ ΙΠΑ κτλ. και να βοηθήσουμε και την Ευρώπη στι εξαγωγέ τη και στην βελτίωση τη ανταγωνιστικότητά τη. Ελπίζω να μα δώσετε κάποιε ειδήσει σε σχέση με την εφαρμογή αυτού του εργαλείου που δεν στοιχίζει, έτσι δεν είναι ακριβό και που θα εκτιμούσε πολύ η βιομηχανία ο κλάδο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα για την ανταγωνιστικότητα και την διαρροή άνθρακα. Όπως είπε και ο κύριος Λίζε, ο οικολογικός σχεδιασμός ε, δρά αντισταθμιστικά για τη διαρροή άνθρακα γιατί ε, εξετάζει με διαφορετικό τρόπο τα εισαγόμενα προϊόντα σχέση με τα ευρωπαϊκά. Και έτσι ενισχύει την ανταγωνιστικότητα γιατί η παραγωγή μας ωφελείται από, τις, ε, ε, από την εξοικονόμηση ενέργεια, γιατί έχουμε και άλλα προϊόντα τα οποία δεν είναι καταναλωτικά, άμεσα καταναλωτικά προϊόντα, απευθύνονται σε άλλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας και στον τομέα το κατασκευαστικό. Για παράδειγμα, αυτή που, ε, επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ανελκυστήρες ή μεγάλα ψυγεία. Η ενεργική εξοικονόμηση βοηθά στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και αυτό ενισχύει την ανταγωνιστικότητα. Δεν θεωρώ ότι η οδηγία οικολογικού σχεδιασμού θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε μορφή διαρροή άνθρακα. Νομίζω ότι μάλλον το αντίθετο σημαίνει. Η επισήμαση, η βιωσιμότητα είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Εξετάζουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη παράδειγμα τη βιωσιμότητα και την ε, αντοχή, ανθεκτικότητα, ε, για να ακολουθήσουμε ε, την οδό που έχουμε ακολουθήσει και στην ενεργειακή επισήμανση. Πρέπει να έχουμε σωστή επισήμανση και να μην εξετάζουμε μόνο κάποιες μερικές λύσεις, γιατί αν κάνουμε τη λάθος επισήμανση, μετά η βιώσιμη κατασκευή και βιομηχανία μπορεί να πληγεί. Αν όμως καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ένα σύστημα όπου οι καταναλωτές να μπορούν να επιλέγουν προϊόντα με βάση την ανθεκτικότητα και όχι μόνο την ενεργειακή απόδοση, νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει την αγορά και θα ενισχύσει και την κυκλική οικονομία. Θα μας βοηθήσει όμως και να μετατρέψουμε ε, γραμμικά επιχειρηματικά μοντέλα για να γίνουν πιο κυκλικά. Ο κύριος Φλόρεντς ρώτησε για το θέμα των ε, απορριμμάτων και αποβλήτων. Δεν είναι έτοιμη η πρότασή μας. Βρισκόμαστε στα πρώιμα στάδια Υπάρχει μια πρωτοβουλία για τη διαπαφή χημικών προϊόντων και της ε, νομοθεσίας ε, περί αποβλήτων. Ε, θέλουμε να ενισχύσουμε την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και των ουσιών στα και στα ανακυκλώσιμα προϊόντα και την εφαρμογή της ταξινόμησης των ευρωπαϊκών προϊόντων. Τέσσερα ζητήματα έχουμε εντοπίσει που παρεμποδίζουν αυτή τη διαδικασία. πρώτα ανεπαρκή ενημέρωση σε, σε ό,τι αφορά τι ουσίε ε, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα προϊόντα και τα απορρίμματα. Μετά, παρουσία ε, προϊόντα και προϊόντων και τέτοιων ουσιών σε ε, ανακυκλώσιμα προϊόντα. Και αβεβαιότητα. για το πώς μπορούν κάποια υλικά να μην θεωρούνται πλέον απορρίμματα και να επαναχρησιμοποιούνται. Βέβαια, αυτό είναι κέρια σημασία ζήτημα όταν εξετάζουμε κίνητρα για την ανακύκλωση ή ευκαιρίες για να διαμορφώσουμε μία ενιαία αγορά για, τα, για τις δευτερογενείς πρωτεσίλες που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Θα επανέλθουμε όμως με μία πρόταση από αυτού στη συνέχεια Τη φετινή χρονιά, όμω προ το πάνω δεν έχω κάτι να πω. Μετά, το θέμα των ηλεκτρικών οχημάτων και τι είδου ε, κίνητρα μπορεί να παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά από την πλευρά των καταναλωτών. Αλλά, για παράδειγμα, υποδομές ε, ε, όπου μπορεί κάποιος να φορτίζει ένα ηλεκτρικό όχημα. Εκεί μπορεί το ΕΦΣΙ να διαδραματίσει ένα ρόλο. Φαντάζομαι λοιπόν ότι μπορούμε να δούμε τι έρχεται πρώτα και όταν τα αυγό. Μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Όταν έχουμε την κρίσιμη μάζα ηλεκτρικών οχημάτων ή όταν φτάσουμε μια κρίσιμη μάζα και πάλι ε, τέτοιων σταθμών ε, ε, φόρτισης, ε, τότε θα μπορούμε να περάσουμε σε μια εποχή με λιγότερες ε, παροχές και επιδοτήσεις. Γιατί συνήθως εμείς αυτό θέλουμε, η αγορά να κινεί τα νήματα και όχι οι δημόσιες επιδοτήσεις. Όμως αυτές οι δύο πηγές χρηματοδότησης ήδη υφίστανται και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τα κρατημέλη να τις αξιοποιήσουν. Κυρία Πιατικάνεν ρώτησε για το ΕΦΣΥ και την κυκλική οικονομία και για δείκτες. Οι δείκτες, όπως έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την αγορά όταν θα ξέρουμε τι είδους δείκτες χρειαζόμαστε και πόσο αξιόπιστοι είναι για τις εκτιμήσεις μας. Όμως, είμαι αρκετά αισιόδοξο, δεν είναι πριν και φυσική. Θεωρητικά τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να είναι. Αλλά προς το παρόν ναι, η Επιτροπή ε, δεν κάνει πολλά σε αυτό το τομέα. Όμως βέβαια στο μέλλον θα τα χρειαστούμε όλα αυτά. Θεωρώ ότι όσο καλύτερη είναι η συνεννόηση και η διαβούλευση μεταξύ και αυτής της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ε, τις ευκαιρίες που μας ε, παρουσιάζονται με τους δείκτες, τόσο καλύτερα θα τα πάμε στο μέλλον. Εύση και κυκλική οικονομία τώρα. Μέχρι τώρα ομολογώ ότι το εύση δεν έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα για, την, για τις επενδύσεις κυκλικής οικονομίας. Δεν γνωρίζω ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό πέρα από τους γνωστού ε, λόγους. Δηλαδή οι επιχειρήσεις που υποτίθεται ότι πρέπει να γνωρίζουν την ύπαρξη και τη λειτουργία του ΕΦΣΥ, ότι δηλαδή μπορεί να χρηματοδοτήσει νέες τεχνολογίες, δεν το γνωρίζουν ε, αρκετά. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε την ε, νομοθεσία που ελπίζουμε να υιοθετηθεί σύντομα για τα απόβλητα και απορρίμματα που θέτει νομικά δεσμευτικούς στόχους για την ανακύκλωση κτλ. Ε, και ασκείται έτσι μεγάλη πίεση ε, για τη δημιουργία νέων τεχνολογιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Έτσι το ΕΦΣΙ μπορεί κάποιος να το δει διαφορετικά στο μέλλον πλέον. Τι άλλο. Καλύτερα να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε την Πρόεδρε που ήρθατε εδώ να τα συζητήσετε όλα αυτά τα ζητήματα του οικολογικού σχεδιασμού μαζί μας όπως ε, ξεκινήσατε κι εσείς και είπατε ότι είναι από τα πιο παρεξηγημένα νομοθετικά πακέτα. Ελπίζω τώρα να τα καταλάβαμε λίγο καλύτερα και θα συνεχίσουμε το διάλογο μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Άρα, uh, συνάδελφοι. Θα κάνω τώρα κάποιες ε, ανακοινώσεις. Συνήθως αυτό έρχεται πρώτο, αλλά ε, ήρθαν αντιπρόεδρος εδώ, οπότε θα κάνουμε τώρα τις ανακοινώσεις που μου ε, προετοίμασε η κυρία Μανιάνα και την ευχαριστώ πολύ, τη γραμματεία. Πρώτον, εφόσον έχουμε την απόφαση τη Ολομέλειας να παραπέμψει και πάλι στην Επιτροπή τον ε, φάκελο τη Ιεκλικής Οικονομίας για ε, διοργανικέ διαπραγματεύσει. και σύμφωνα και με τον κανόνα 69, η ομάδα διαπραγμάτευση ε, ε, τη ομάδα μάλλον θα προεδρεύσει η πρόεδρο και βέβαια θα συμμετάσχουν ε, ο εισηγητή και οι σκιώδει ω συνήθω. Δεύτερον, εφόσον έχουμε κάποια προβλήματα με την ε, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών που είναι στις 12, από ό,τι φαίνεται οι επιτροπές λάμπαναν μία ακριβή ώρα ως προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για να κατατίθενται όλες ε, έτσι. Δεν είναι πολιτική απόφαση βέβαια αυτό, είναι πιο τυπικό το ζήτημα. Από τούτο και στο εξή, για την Επιτροπή μας, οι τροπολογίε θα κατατίθενται έως τις 11. Βέβαια, όπως είπα και στους συντονιστέ, επαναλαμβάνω ότι αν υπάρχει κάτι κατεπήγον, μπορείτε να ζητήσετε να κατατεθεί και στη συνέχεια και σίγουρα θα σας βοηθήσει και η γραμματεία να καταθέσετε τροπολογίες και μετά τις 11. Στο ίντρανετ τώρα έχουμε ένα νέο τμήμα για σας όπου μπορείτε να βρείτε καταξιδότηση και εκτελεστικές πράξεις βέβαια που άφτονται των ε, δικών μας ε, θεμάτων. Βέβαια, χρειάζεστε και τις οδηγίες της γραμματείας για να ε, έχετε πρόσβαση εκεί. Θα, στείλει μέσω, θα σταλεί μέσω mail στα μέλη μας και στους συμβούλους των πολιτικών ομάδων. Μετά, υπερθυμίζω ότι έχουμε μία ακρόαση της Γιούρη της ε, στις 11 Απριλίου στις 3.30 ε, στο πλαίσιο της ε, συνεδρίας της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Καλό είναι λοιπόν να ενθαρρύνετε και τους συναδέλφους μας να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Μετά, στο φάκελό σας έχετε και την έκθεση για την αποστολή προς τον Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Οργανισμό που έλαβε χώρα τον Νοέμβρη, τη οποία ηγήθηκε ο κύριο Σουαρία και αν θέλετε να ενημερωθείτε για την αποστολή αυτή θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο φάκελό σα. Μετά, λυπούμε να σα ενημερώσω ότι ο κύριος Γιώργος Αμανατίδης, σημαντικό μέλο ε, της ε, ομάδας μας, ε, θα αποχωρήσει από την γραμματεία της ΕΝΒΗ, όχι επειδή το επιθυμούμε, αλλά στο πλαίσιο της ε, εκπεριτροπής ανάληψης θέσεων ε, ε, του Κοινοβουλίου θα πάει στο Τμήμα Πολιτικής Α και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας ε, και κατά αυτόν τον τρόπο σας εύχομαι καλή επιτυχία και να σας πω ότι εκτιμήσαμε πολύ την παρουσία σας στη Γραμματεία και θα μας λείψετε. Uh, Αυτές ήταν οι πιο σημαντικές ε, ανακοινώσεις της Προέδρου. Έχουμε τερμηνία σε 21 γλώσσες και βεβαίως ε, η συνεδρίαση μεταδίδεται και μέσω διαδικτύου. Στους φακέλους σας θα βρείτε και τα πρακτικά της ε, συνεδρίασης της 23ης και 24ης Ιανουαρίου. Επειδή τα πρακτικά μεταφράζονται σε πολλές γλώσσες, ε, καθυστερεί ε, η τελική τους έγκριση. Μπορούμε να το εξετάσουμε και στα, στους συντονιστές. Τέλος πάντων, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις και αντιρρήσεις προς τα πρακτικά, θεωρώ ότι εγκρίνονται. Αυτά σε ό,τι αφορά τα, τις ανακοινώσεις Προέδρου και μπορούμε τώρα να περάσουμε στα πιο ουσιώδη για μας. Πρώτον έχουμε το σχέδιο κανονισμού δεύτερης ανάγνωσης για την έκθεση της κυρίας Βίλμοντ ε, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα να σας αναφέρω το χρονοδιάγραμμα. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΝΒΙ αύριο και μετά στην Ολομέλεια την 1η Απριλίου. Το ίδιο χρονοδιάγραμμα ισχύει και για τα in vitro διαγνωστικά για τεχνολογικά προϊόντα, την έκθεση του κ. Λίζα. Όχι, για το επόμενο θέμα δεν ισχύει το ίδιο διάγραμμα. Θα πρέπει να περιμένουμε τη δεύτερη ανάγνωση. Ας περάσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα που είναι το σχέδιο σύσταση σε ό,τι αφορά τη σύμβαση της Μιναμάτα για τον Ιδράργυρο. Το λόγο έχει ο εισηγητής κύριος Στέφαν Εκ. Yeah, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τι υπάρχει άλλο να πούμε, πέρα από αυτό που ψηφίσαμε την τελευταία εβδομάδα στην Ολομέλεια. Ε, να πω πως χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η έκθεση δεδομένη της χρονικής πίεσης ε, καταφέραμε να ψηφιστεί τόσο γρήγορα. Παρότι υπήρχαν κάποια σημεία στην έκθεση τα οποία θα ευχόμουν ένα πιο φιλόδοξα. Όμως το σημαντικό είναι ότι με αυτή τη σύμβαση της Μιναμάτα καταφέραμε να αποκτήσουμε στο μέλλον τη δυνατότητα να πάμε ένα βήμα προς ε, την ε, σταδιακή εξάλληψη του υδραργύρου. Περνάμε σε μία ακόμα μείωση. Όλοι γνωρίζουμε πόσο τοξικός είναι ο υδράργυρος και πόσο γρήγορα γίνεται τοξικός. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να χαιρετήσω την ταχύτητα με την οποία εργαστήκαμε, να πω ότι στη Γενέβη θα, το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, θα ε, ε, γίνει ένα συνέδριο για τη σύμβαση της Μιναμάτα και ε, πρέπει να ασκήσουμε την κατάλληλη πίεση έτσι ώστε στο μέλλον να είμαστε ακόμα πιο φιλόδοξοι, ακόμα πιο εργατικοί έτσι ώστε να μειωθεί ακόμα περισσότερο ε, η χρήση του υδράργυρου σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς. Και ε, οι περιοχές που έχουν μολυνθεί από διάφορες διαρροές υδραργύρου ε, να ε, προσπαθήσουμε να καθαριστούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος ε, που καταφέραμε και ψηφίσαμε αυτή την έκθεση και περιμένω με αγωνία να δω τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους και εισηγητές. Εκ μέρους λοιπόν του ΕΛΚ ε, θα ήθελε κάποιος να λάβει το λόγο. Ο κύριος Νταντέν που είναι σχεδόν ηγητής λείπει από ό,τι βλέπω. Βλείπει ε, και ο κύριος Παουλούτσι ή δεν τον βλέπω εγώ. Θα τον αντικαταστήσει κάποιος. Κύριε Ντάλη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Παουλούτσι δεν κατάφερε να έρθει όμως ε, μου έστειλε ένα σημείωμα με δύο λόγια που θα ήθελα να σας μεταφέρω. Είναι λοιπόν πολύ ικανοποιημένο που η Ολομέλεια ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία την προσωρινή συμφωνία για τον κανονισμό περί υδραργύρου που θα τεθεί σύντομα σε ισχύ και θα εφαρμόσει τις αποφάσεις της ε, Σύμβασης της Μιναμάτα. Είναι η πρώτη παγκόσμια δεσμευτική συμφωνία ε, για τον υδράργυρο. με ένα από τα πιο μία από τις πιο τοξικές ε, ουσίες. Είναι λοιπόν ε, καιρός να προχωρήσουμε ως το δυνατόν γρηγορότερα στην κύρωση της ίδιας της συμφωνίας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέρος ε, στην πρώτη συνάντηση τον Σεπτέμβριο, 20 Σεπτεμβρίου, στη Γενέβη για τη Σύμβαση της Μιναμάτα και να συζητηθούν οι λεπτομέρειες σχετικά. Γι' αυτό λοιπόν θα υποστηρίξουμε ε, την ε, ε, έκθεση με την ψηφοφορία αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου τη ομάδα CCR δεν υπάρχει κάποιο. Φιλελεύθερη. Πράσινη. Κύριο Πιδιτσίνη, λείπει. Κύριε κυρία Τορνάνο έφυγε. Τώρα λοιπόν, όποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο, παρακαλώ να το ζητήσει. Κανείς. Μάλιστα, φαίνεται πως είμαστε όλοι σαφείς και σύμφωνοι. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Η Κομισιόν καλωσορίζει τις συστάσεις του εισηγητή, κυρίου ΕΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρέχει τη συγκατάθεσή του για την ε, κύρωση της συμφωνίας της Μιναμάτα για τον Ιδράργυρο η επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα διασφαλίσει την γρήγορη θέση ισχύ της σύμβασης και τις ε, γρήγορες και άμεσες κυρώσεις σε όσους ρηπαίνουν με υδράργυρο. Αυτό θα ωφελήσει σημαντικά τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς το 48% των, ε, του υδραργύρου που εκλείεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παράγεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγεται. Προγραμματίζεται λοιπόν ε, η πρώτη συνάντηση στα τέλη Σεπτεμβρίου, γι' αυτό λοιπόν η επικύρωση πρέπει να γίνει πριν τα τέλη Ιουνίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει απόλυτα ότι πρέπει όλα τα κρατημέλη να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επικύρωσης μέχρι τότε, όμως δεν πρέπει να υπάρχουν καθυστερήσεις ε, που με τη σειρά τους θα καθυστερήσουν την ε, σε ισχύ τη ε, σύμβαση της Μιναμάτα. Πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο ε, μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να είναι πρωτοπόρος ε, στην προσπάθεια εξάλληψης του υδραργύρου από την οικονομία. Αυτό πιστεύω θα δώσει και το καλό παράδειγμα στους διεθνείς μας εταίρους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα ξανά αν υπάρχει κάποιος από εσάς που θέλει να λάβει το λόγο για αυτό το θέμα της ενέργειας διάταξης, τη σύμβαση της Μιναμάτα. Όχι. Ο λόγος πίσω σε εσάς, κύριε Εκ. Κύριε Εκ, με συγχωρείτε, ε, έχει να κάνει με την αντίρρηση για τα μεταλλαγμένα. Όχι, εντάξει, συγγνώμη. Όχι, Μιναμάτα, το είπα. Το είπα μόλις. Σύμβαση της Μιναμάτα. Δεν ακούσατε στο προηγούμενο σημείο είμαστε ακόμα. Ε, κύριε Εκ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Βλέπω πως δυστυχώς δεν είχαμε πολλές τοποθετήσεις σε αυτό το θέμα, αλλά θα μπορούσε κανείς να το δει ε, και αλλιώς, ότι δηλαδή όλοι συμφωνούμε. Και Συμφωνούμε και για το περιεχόμενο της έκθεσης και για την γρήγορη επικύρωση της σύμβασης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να επικυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη σύμβαση και να έχει πρωτοπόρο ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες μείωσης ε, του υδραργύρου. Πρέπει λοιπόν από την Ευρώπη να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι εμείς παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά την περιβαλλοντική πολιτική. Ακριβώς διότι η περιβαλλοντική πολιτική είναι και κοινωνική πολιτική. Και είναι γι' αυτό αναγκαίο η κοινωνία να ε, αποκτήσει πλήρη αντίληψη ε, του πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα, πόσα ευθύνη έχει για την υγεία ε, των ανθρώπων, την υγεία των ζώων και την υγεία όλου του πλανήτη. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ, ξαναλέω, που στην Ολομέλεια ψηφίστηκε με τόσο μεγάλη πλειοψηφία η έκθεση και ελπίζω το μέλλον να μας επιφυλάξει θετικές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε βαζή θα θέλατε να πείτε κάτι. Έχετε το λόγο αν θέλετε. Ναι. Σχετικά με το κείμενο που ψηφίσαμε 17 Μαρτίου στο Κοινοβούλιο να θέσω ένα ερώτημα για την επικύρωση αυτής της σύμβασης μηναματά. Ξέρετε ότι 26 χώρες έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν επικυρώσει την μηναμάτα για τον Ιδράργυρο. Είπε την Αιγύρια του προγράμματος του ΙΕ για το περιβάλλον που υιοθετήθηκε το 2013. 120 έχουν υπογράψει, 38 μόνο έχουν επικυρώσει. Κίνα, ΙΠΑ, σημερινό κτλ. Χρειάζεται λοιπόν η επικύρωση 50 χωρών για να τεθεί σε ισχύ 24 ώρες μετά από την υπογραφή της επικύρωσης. Για το Σεπτέμβριο λοιπόν, στη Γενέβη προβλέπεται αυτή. Θέλουμε λοιπόν η Ευρώπη και η ΕΠΑ να επικυρώσουν την σύμβαση αυτή πριν αυτή την ημερομηνία, πριν το Σεπτέμβριο, ώστε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Η Ευρώπη λοιπόν να επικυρώσει αυτή την σύμβαση όπως και οι χώρες μέλη της. Και αν γίνεται πριν από την ΚΟΠ της Γενέβης. Αυτό θα ήταν πολύ ισχυρό μήνυμα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Μια και ήρθε ο κύριος Σκιώδης του Αλεξάντα. Έχετε το λόγο. Ήμουν σε άλλη επιτροπή για παρόμοιο θέμα, Πρόεδρε. Η επικύρωση της Μιναμάτα του Γενάρη του 2013 αποτελεί μια εργασία με την οποία ασχολούμαστε εδώ και ένα χρόνο για την καταπολέμηση των βλαβερών συνεπειών του Ιδράργυρου. Νομίζω ότι έχουμε ένα φιλόδοξο και ελιστικό κείμενο και χαιρόμαστε γι' αυτό με κανόνες που ευθυγραμμίζουν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο με το πρόγραμμα του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του υδραργύρου. Νομίζω θα πρέπει να συνεχίσουμε να αποτελούμε ένα παράδειγμα και η ταχεία επικύρωση θα μας επιτρέψει ακριβώς στην Ένωση σε όλους μας να παίξει ένα ρόλο κινητήριας δύναμης το Σεπτέμβρη στην Κόπτη, στη Γενέβη. Έχουμε εργαστεί με καθυστερήσεις παλαιότερα. Οπότε τώρα νομίζω θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Ό,τι μπορούμε και ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ. Επιτροπή Κομισιόν θέλετε να σχολιάσετε αυτά τα σχόλια. Ξέρω ότι εντάξει ξαναμιλήσατε αλλά ναι για τις φάσεις της επικύρωσης χρειαζόταν η επικύρωση τη ΕΕ πριν σε επικύρωση των χωρών μελών. Αλλά ήδη αρκετέ χώρε ήταν έτοιμε γι' αυτό, για τη δικιά του δηλαδή διαδικασία. Οπότε έχουμε 38, χρειαζόμαστε άλλε 12, ώστε να τεθεί σε ισχύ η σύμβαση. Ξέρουμε ότι 6 χώρε ήδη είναι έτοιμε για την επικύρωση και από επαφές που είχαμε με χώρες μέλη Άλλες 6-7 χώρες μας είπαν θα είναι έτοιμες έγκυρα για να επικυρώσει και η Ένωση. Ελπίζουμε λοιπόν η επικύρωση της Ένωσης να προκαλέσει την θέση ισχύ τη σύμβασης ώστε αυτό να αποτελέσει τέλο πάντων μεγάλη διαφήμιση για την ΕΕ όσον αφορά τη διάσωση των πολιτών του κόσμου όσον αφορά τις φλαβερές συνέπειε των εκπομπών δραγύρου. Ευχαριστώ και καλή τύχη, λέει πρόεδρο. Εκ, θέλετε το λόγο. Όχι, δεν θέλετε. Α, καλά, τότε, τότε εντάξει. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σα. Τελειώσαμε αυτό το σημείο 7 λοιπόν για τον Ενδράργυρο και την Μίνα Μάτα. Οπότε προχωράμε. Uh, Επόμενο σημείο στη μερίσια μας γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Δικατοέξι. Δικασία. Αντίσταση αφορά το 106. Πρόεδρο γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου συγκεκριμένα. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο για το σχέδιο ψηφίσματος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ακόμα μερικούς συναδέλφους, ε, πράγματι, ε, κάναμε μια πρόταση αντίρρησης ό,τι αφορά την έγκριση ε, αυτού του τύπου αραβοσίτου Όποιος διαβάσει καλά το έγγραφο καταλαβαίνει ότι ο σκοπός ε, αυτής της, ε, αυτού του αιτήματος της Συγγέντα και ε, η σύσταση να δοθεί αδειοδότηση από την Επιτροπή είναι η αποτροπή διάφορων ασθενειών για τον αραβόσιτο αλλά πρόκειται και για ουσίες που περιλαμβάνουν και γλυφοσάτ και άλλες βλαβερές ουσίες. Υπάρχει μια γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ του 2016 και βλέπουμε ότι πρόκειται όντω για θετική γνωμοδότηση. Όμω, αν την εξετάσει κανεί με προσοχή, βλέπουμε ότι υπάρχει και μία, ή πρόκειται για μία γνωμοδότηση ε, μειοψηφία εντό ε, τη ΕΦΣΑ. Όμω προτείνεται να εγκριθεί γιατί η Συνγέντα έχει κάνει το αρχικό αίτημα αλλά έχει διευρύνει αυτό το αίτημα και σε μία σειρά περίπου 20 υποσυνδυασμών. Όμως εκεί ε, σημαντικός αριθμός αυτών των ε, υποσυνδυασμών ε, μη γενετικά τροποποιημένων οργανισμών δεν υπάρχουν καν, οπότε δεν έχει γίνει ο, έλεγχος για το κατά είναι ασφαλής. και δεν υπάρχει επαρκής επιστημονική βιβλιογραφία. Παρ' όλα αυτά, η ΕΦΣΑ λέει ότι αυτές οι 20 υποενώσεις είναι εξίσου ασφαλείς ε, όσο ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός με τα 5 υποτμήματα. Με τη διαβούλευση με τα πέντε κράτη-μέλη βλέπουμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες επικριτικές παρατηρήσεις από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά ε, την έλλειψη στοιχείων, μελετών, βιβλιογραφίας, ε, στοιχείων σε ό,τι αφορά το, σχετικά με το συνδυασμό των επιπτώσεων, ε, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των field tests ε, σε ό,τι αφορά την επίπτωση αυτού του οργανισμού ε, στο περιβάλλον. Η έκθεση μειοψηφία, λοιπόν, η σύσταση μειοψηφία του κυρίου Βαλ λέει ότι για αυτούς τους 20 υποσυνδυασμούς δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Η Συγγέντα ε, δεν έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις γιατί, δεν γιατί δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Μπορείτε να διαβάσετε όλα αυτά τα στοιχεία στο σχέδιο ψηφίσματος ε, που θα καταθέσουμε αύριο ε, στις τελικέ σκέψεις J, K και L. Υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση ό,τι αφορά την ε, αντοχή, σε ό,τι αφορά το γλυφοσινάτ, υπάρχει και το γλυφοσάτ και το όριο δηλαδή το επιτρεπόμενο. Ξέρετε ότι αυτή η συζήτηση ακόμα συνεχίζεται και μετά την ε, έκθεση της ΕΤΣΑ την περασμένη εβδομάδα και σε όλο αυτό το πλαίσιο λαμβάνουμε υπόψη και τη διαδικασία. Η μόνιμη Διαρκής Επιτροπή των κρατών, κρατών Μελών έχει ήδη κάνει μια πρώτη συνάντηση και βλέπουμε ότι μόλις 10 από τα 28 κράτη-μέλη στηρίζουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσωπούν μόλις το 38% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Γι' αυτό έχουμε καταθέσει με τους συναδέλφους αυτή την ε, ε, ένσταση τα επιχειρήματά μας ε, τα έχουμε συλλέξει και σε ένα ψήφισμα το οποίο θα ε, ψηφίσουμε αύριο. Εκεί υπάρχουν όλα τα επιχειρήματα ε, και γι' αυτό καλώ και του συναδέλφους να στηρίξουν αυτή την ένσταση. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να δώσουμε το λόγο στους σκιώδεις, μάλλον συνεισηγητές. Αν είναι κανείς εδώ, αν θέλει να πάρει το λόγο. Κανείς? Όχι. Μετά, σκιώδης. Η κυρία Γιουσο. παρακαλώ. Πρώτα ευχαριστώ. Εξ ονόματος του ΕΛΚ πρέπει να πω ότι όπως είπε σωστά ο συγητής έχουμε να κάνουμε ένα γενετικά τροπευμένο τύπο αναποσίτου και αφορά συγκεκριμένα στοιχεία και συστατικά τροφίμων που έχουν παραχθεί ή παρασκευαστεί με τον αγώστο αυτό και αφορούν και την καλλιεργία του. Εδώ έχουμε κάνει μια εκτελεστική πράξη. Οπότε πρέπει να είμαστε συνεπείς και να πούμε ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλο ένα παράδειγμα κατάχρησης στο Κοινοβούλιο σε σχέση με αυτές τις εκκληστικές πράξεις. Για την ΕΦΣΑ, να πω σε συγκεκριμένα πέντε παραγράφους που αφορά αυτό και τη μειοψηφική άποψη των διαφόρων εμπειρογνωμόνων. Είχαμε στην ΕΦΣΑ μια διαδικασία αξιολόγησης. Όταν έγινε αυτή η αξιολόγηση, και η γνωμοδότηση μειο, μειοψηφία δεν σημαίνει ότι είχαμε, είχαμε βασιστεί σε συγκεκριμένα γεγονότα. Όπως είπαμε, δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επειδή μας αρέσουν. Και η ΕΦΣΑ είχε ταχθεί υπέρ, τα θετική. Να πω επίσης για την γλυφοσάτη, αυτά που ακούσαμε προηγουμένως, δεν έχουν νόημα γιατί δεν αφορούν την καλλιέργεια του αραβόσιτου αλλά την χρήση του στην παρασκευή συγκεκριμένων τροφίμων. Οπότε η, το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την γλυφωσάτη από τη στιγμή που έχουμε καλλιέργεια νομίζω ότι αυτό δεν στέκει και εμείς θα καταψηφίσουμε ανεξάρτητα βέβαια το γεγονό ότι θα υπάρξουν κάποια μέλη τη πολιτική μα ομάδα που έχουν δική του άποψη διαφορετική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γαβοστέτ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με την κυρία Γιούσο και θα αναφερθώ σε αυτά που έθιξε. Δεκάδες φορές έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Επομένω, θα σταθώ περισσότερο στο ε, πρόβλημα του τύπου και έχει τόσο στην ουσία, γιατί εκεί συμφωνώ με την κυρία Γιούσο διαρωτώ με και ανησυχώ σε ό,τι αφορά ε, τον πολλαπλασιασμό αυτών των ε, κατεξοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που μας ε, υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, δεν έχουμε πάντα και εμείς και τα κρατη δυνατότητα να τα ελέγξουμε. Σε ό,τι αφορά τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς πρόκειται για συνήθεις διαδικασίες βάσει ανάλυση κινδύνου και ερευνών που γίνεται από την ΕΦΣΑ. Πολλές φορές αυτές οι ενστάσεις ε, ε, οδηγούν ε, σε έναν πολιτικό αντιπερισπασμό για να διαμορφώσουν πολύ μεγαλύτερο όγκο εργασιών στις επιτροπές. Και η Επιτροπή μας έτσι χάνει απολύτως την αξιοπιστία της. Σε ό,τι αφορά ε, την αδειοδότηση των ε, ε, γάμματα αφόμικρων έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο γίνεται σεβαστό γενικά βάσει και της ανάλυσης κινδύνου που γίνεται από τον οργανισμό μας, την ΕΦΣΑ. Επομένω, καλό θα ήταν επιτέλου ε, να σταματήσουμε να αμφισβητούμε αυτή τη διαδικασία. Και να, με το να κάνουμε συνεχώ ε, ε, και ακατάπαυστα ενστάσει βάσει του άρθρου 106, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάχρησης της διαδικασίας. Και εδώ αναφέρομαι στο, στο άρθρο 106 παράγραφος 2 του κανονισμού που αναφέρει ότι η αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει στο Κοινοβούλιο ένα σχέδιο ε, ψηφίσματος που αναφέρει ότι ένα σχέδιο, μια πρόταση εκτελεστικού ε, μέτρου ε, υπερβαίνει τι αρμοδιότητε ή δεν συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο για άλλου λόγου. Και όταν έχουμε λοιπόν ε, και για αυτού του δύο λόγου. Ε, έχουμε λοιπόν την ένσταση. Αλλά κανένα από αυτά τα δύο στοιχεία δεν υπάρχει εμπροκειμένο. Επομένω, δεν υπάρχει λόγο ύπαρξη αυτή τη ένσταση. Και νομίζω ότι η Επιτροπή μου θα πρέπει. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να ε, διαμορφώσει ένα πλαίσιο και να συμμορφούνται με αυτές ε, τις διατάξεις, με αυτούς τους κανόνες, όπως ισχύει και για άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, γιατί αυτό θα βοηθήσει ε, τη λειτουργία της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκροστέτ, συμφωνώ και εγώ μαζί σας απόλυτα. Πρέπει να δώσουμε τη δέουσα σημασία σε αυτές τις ενστάσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες. Και πολλές φορές ε, το περισσότερο σημαίνει λιγότερο. Είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί στους συντονιστές Γι' αυτό λοιπόν ε, μεταφέρετε το στους συναδέλφους σας και ας δούμε πώς μπορούμε ε, από εδώ και στο εξής να χειριζόμαστε καλύτερα παρόμοια θέματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ ε, και τώρα δώσω το λόγο στον κύριο Πανιά. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή ευκαιρία τώρα αυτή η συζήτηση, γιατί εγώ διαφωνώ. Σκέφτομαι ακριβώ το αντίθετο από αυτό που άκουσα. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα και το να λέει κανεί ότι ε, το, το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα με τι αρμοδιότητέ του να εκφέρει γνώμη σε μια τέτοια διαδικασία και με τι δυνατότητε τη ένσταση, για μένα όχι απλά είναι κάτι το χρήσιμο, αλλά είναι και ένα μέσο προστασία ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί πολύ συχνά εδώ ε, λυπούμεθα για την κακή εικόνα που έχουν οι Ευρωπαίοι συμπολίτε μα. Όμω κάποιε φορέ αυτό είναι γιατί δεν είχαμε το κουράγιο και το θάρρο να καταδείξουμε τα κακό ακόμα και αν δυσαρεστήσουμε ε, τη βιομηχανία και έτσι να βελτιώσουμε όμως και την εικόνα των θεσμικών οργάνων και να μην είναι μόνο οι αντιευρωπαϊστές και οι εθνικιστές ε, που θα ακούγονται κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών εκλογών όπως είδαμε δυστυχώς το 2014. Όμως ε, ε, παίρνω το λόγο σήμερα εξ ονόματος του συναδέλφου Μπαλάς που δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα γιατί συνεχίζει την προεδρική προεκλογική εκστρατεία. Όπως ξέρετε, κ. Μπαλά με μια σειρά ευρωβουλευτών από πολλές πολιτικές ομάδες ε, ε, παρακολουθούν τις διαδικασίες ε, στα της επιτροπολογίας για να παρακολουθούν τις διαδικασίες για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Εδώ πρόκειται για μια αντίρρηση στην ε, έγκριση εκτελεστικής πράξης για 28 διαφορετικά προϊόντα σε συγκεκριμένε κατηγορίες ε, και ποικιλίε αραβοσίτου που θα είναι ανθεκτικά στα ζενιοκτώνα, γλυφοσινάτ, γλυφοσάτ, και άλλες ουσίες. Η Συνζέντα λοιπόν την 1η Ιουλίου του 2011 κατέθεσε έτοιμα ε, κυκλοφορίας, εμπορίας συγκεκριμένων ε, ζωοτροφών και άλλων ε, υλικών για μια σειρά διαφορετικών γενετικών τροποποιημένων γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών. Πρέπει να είμαστε ακριβεί και αυτό κάνουμε και εμεί εδώ. Γιατί μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα η υγεία και η επιστημιακή ασφάλεια. Δεν θεωρούμε ότι είναι καλό να υιοθετήσουμε και να εγκρίνουμε ε, τέτοιε ποικιλίε που δεν έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί. Πρόκειται για μια έκθεση μειοψηφία λοιπόν που δεν αναφέρει κανένα συγκεκριμένο στοιχείο σε ό,τι αφορά αυτούς τους 20 υποσυνδυασμούς που έχει ε, δώσει η Συντζέντα και ούτε έχει δώσει η ίδια η εταιρεία επαρκής ε, αιτιολογήσεις ε, για αυτά τα στοιχεία και γιατί θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη αυτά τα στοιχεία που λείπουν για την αξιολόγηση δικτύπου. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δεν είναι εδώ ο κύριος Μπάλας, οπότε δεν μπορούμε να του δώσουμε και περισσότερο χρόνο. Καταλαβαίνετε. Ε, άλλα μέλη που θέλω να πάρουν το λόγο. Τρία μέλη. Κυρία Πιατικάινεν, παρακαλώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Δύο ειδών κίνδυνοι υπάρχουν στη ζωή μας. Οι εύκολοι και αυτοί που είναι αναστρέψιμοι. Δηλαδή, αν ε, πέσω μπροστά σε ένα αυτοκίνητο, μπορεί να, θα χτυπήσω, αλλά και κάποιος μπορεί μετά να ε, με επαναφέρει. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι κίνδυνοι, οι μη αναστρέψιμοι, που είναι ιδιαίτερα ε, βλαβαροί, καταστροφικοί και κίνδυνοι για τους οποίους δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και θα ήθελα λοιπόν να σας παροτρύνω να διαβάσετε το Black Swan του Nassim Τάλετ. Είναι ένας από τους πιο έγκριτους ερευνητές τις μέρες μας. Και ασχολείται με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, με, τα, με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, με την πυρηνική ενέργεια κτλ. Είναι μια μεγάλη αλυσίδα ε, και αναφέρεται σε αυτές τις ουσίες οι οποίες ε, έχουν μακροχρόνιες ε, βλαβαρές επιπτώσεις στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες αρχές, προληπτικές αρχές ε, σε παγκόσμιο επίπεδο για πολλά θέματα, για την πυρηνική ενέργεια για παράδειγμα, όπως ακούσαμε πριν τον υδράργυρο κτλ. Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί δεν μας ε, σκοτώνουν άμεσα, όμως η, επιδράση, η επίδραση τους ε, γίνεται μακροπρόθεσμα. Και εδώ πιστεύω πως έχει γίνει ένα μεγάλο λάθος. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σημαντικό το θέμα αυτό. Δεν έχει να κάνει με ένα τεχνικό ζήτημα, με το τι είναι περισσότερο, τι είναι υπερβολικό, τι πρέπει να γίνει ε, κτλ. Να το πω διαφορετικά. Ε, ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ε, δώσει υπερβολικά πολλές εγκρίσεις για τέτοιους οργανισμούς και κάτι που δεν θα έπρεπε πιστεύω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξέρετε, υπάρχουν κανόνε, υπάρχει κανονισμό για όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, μπορούμε να διαβάσουμε, να μορφωθούμε, όπω είπατε. Δεν λέω βέβαια πω αυτά που λέτε είναι ασήμαντα, κάθε άλλο. Αλλά πρέπει να ακολουθούμε τους, ε, τον κανονισμό. Η κυρία Γκέρλινγκ τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Να επιστήσω, αγαπητοί συνάδελφοι, την προσοχή σα στο ότι σύμφωνα με τον κανονισμό περί επιτροπολογία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει ένσταση μόνο όταν η Κομισιόν υπερβαίνει των αρμοδιοτήτων τη, των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων τη. Γι' αυτό λοιπόν η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση αυτή δεν το έχει κάνει. Δεν έχει υπερβεί τι εκτελεστικέ τη αρμοδιότητε σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Δεν βλέπω κάποια απόδειξη για το αντίθετο προσωπικά και να αναφέρω ότι κάθε φορά που γίνονται ενστάσεις για ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, βλέπω ε, πώς ε, γίνεται η ίδια ιστορία. Γιατί ασκούμε ενστάσεις χωρίς υπόβαθρο, χωρίς κάποια στοιχεία. Υπάρχει μία μειοψηφία η οποία το κάνει αυτό, να το τονίσουμε αυτό, μειοψηφία και η επιστημονική ομάδα που κάνει αυτούς τους ισχυρισμούς δεν είναι... Δεν ανήκει στην πλειοψηφία. Να το τονίσω αυτό. Η πλειοψηφία έχει διαφορετική άποψη. Τώρα, σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφαση, δώσαμε αυτή την εντολή στην ΕΦΣΑ, δώσαμε εκτελεστικέ αρμοδιότητε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα, εάν φτάσουμε στο σημείο να τα αμφισβητούμε αυτά, τότε να αμφισβητήσουμε τα πάντα. Να αμφισβητήσουμε όλε τι εκτελεστικέ πράξει. Αυτό είναι ένα ε, πολύ επικίνδυνο μονοπάτι που διαβαίνουμε. Υπάρχουν ε, αυτές οι ανεξάρτητες ε, μελέτες ε, επιπτώσεων και πρέπει αυτές ε, να, τις, να τους δώσουμε την βαρύτητα που τους αρμόζει. Τώρα, θα ήθελα επίσης να σας επιστήσω την προσοχή στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Τι σημαίνει μια αναστρέψιμες βλάβης. Ε, δεν είναι κάτι που θα μας σκοτώσει αμέσως, είπατε. Είναι απίστευτα αυτά που ακούω. Μας είπατε ότι θα μας σκοτώσει κάποια στιγμή αυτό. Είναι μία αναστρέψιμο. Δεν υπάρχουν αποδείξεις, δεν υπάρχουν στοιχεία για το ότι ε, τα γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ε, θα ε, είναι θανατηφόροι. Όχι, αυτή είναι η ισχυρισμοί σας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκέρλιν, ε, κυρία Ρίβας έχει το λόγο. Παρακαλώ συνεχίστε διμερώς τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Παραξενεύομαι που αφισβητούμε αυτές τις αντιρρήσεις. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με τα καθήκοντα και τις εξουσίες των βουλευτών. Αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα μπορούσαμε να αφισβητήσουμε αυτά που κάνει η Κομισιόν με την καλλιέργεια αυτών των οργανισμών, των τροπομεμένων, όπως έφεραν και άλλοι συνάδελφοι. Και το γεγονό ότι ο ΕΦΣΑ γνωμοδότησε θετικά. Ξέρετε τι γίνεται με τον ΕΦΣΑ. Υπάρχει μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων. Είδατε τι έγινε με την γλυφοσάτη. Δεν μα έδωσαν τι μελέτε. Και το μαρτυρό, το καταμαρτυρό αυτό, μα έδωσαν μελέτε για την γλυφοσάτη που δεν έγιναν ε, έτσι, γνωστές, δεν δημοσιοποιήθηκαν. Δεν γίνεται λοιπόν με αυτή την κατάσταση να συνεχίσουμε. Να σκεφτούμε λοιπόν Ποιος είναι ο λόγος να έχει κανείς έκριση για τροποποιημένους οργανισμούς που αντιστέκονται, που είναι θεκτικοί στο, στην γλυφωσάτη, τη στιγμή που έχουμε non-paper, τα οποία τέλος πάντων μιλούν για γεωργού, για ε, καρκίνο κλπ. κλπ. Είχαμε ποικιλίε οι οποίες ε, βγήκαν από, τις, από την ταξινόμηση. Ο James Περίο, ο μεγάλος ειδικό για την γλυφοσάτη, με 300 σκευάλια δημοσιεύσεις, είχε πει ότι η γλυφοσάτη προκαλούσε μεταλλάξεις. Η Μονσάτο λοιπόν έκανε τα πάντα ώστε αυτός ο μεγάλος επιστήμονας να δώσει διαφορετική άποψη. Και αυτός αρνήθηκε. Η επιστήμη του, η επιστημοσύνη του λοιπόν βασίζεται σε μελέτες. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτό που δήλωσε η ΕΦΣΑ και η ΕΚΑ. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με κάτι το οποίο ενοχλεί τέλο πάντων, προκαλεί βλάβε, αλλά είναι καρκινογόνο και μεταλλαξιογόνο. Ε, επιτρέψτε μου λοιπόν να διατυπώσω αμφιβολίες σε σχέση με τις νομοδοτήσεις της ΕΦΣΑ. Και δεύτερον, γιατί χρειαζόμαστε τι αντιρρήσει αυτέ. Χρειαζόμαστε τι αντιρρήσει αυτέ επειδή συμφωνούν όλε οι χώρε μέλη. Κοιτάξτε τι έγινε στην προηγούμενη συνάντηση τη ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Δέκα χώρε ήταν έτοιμε να υπερψηφίσουν, αλλά 13 χώρε ήταν κατά τη αδειοδότηση. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο λοιπόν θέση των βουλευτών, αλλά με τη θέση πολλών χωρών μελών. Δεν θέλουμε του ε, οργανισμού που είναι ανθεκτικοί στην γλυφοσάτη, γιατί κατά πάσα πιθανότητα η είναι καρκινογόνο, οπότε δεν έχει νόημα τα κάνουμε όλα αυτά. Παρακαλώ να ακολουθήσετε το χρόνο μιλία ε, των δύο λεπτών ώστε να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Λέει η Πρόεδρο. Μήπω κάποιο άλλο θα ήθελε το λόγο. Κύριε Γκροστέτ και πάλι. Όχι. Ε, λυπάμαι. το κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για τόσο ευαίσθητα θέματα όπως αυτοί οι οργανισμοί. Θα ήθελα όμως να είμαστε λογικοί εδώ. Χάρη στους οργανισμούς αυτούς έχουμε βρει κάποια φάρμακα τα οποία είναι απαραίτητα. Δεν χρειάζεται συστηματικά να καταδικάζουμε όλους τους γενικά τροπομένους οργανισμούς. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Όταν θα πρέπει να θρέψουμε δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη, δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό χωρίς τους γενικά τροπομένους οργανισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κάποιος άλλος. Επιθυμεί το λόγο, λέει η πρόεδρος. Όχι, η Κομισιόν τότε. Όχι ούτε η Κομισιόν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο. Ακούσαμε βεβαίως με μεγάλο ενδιαφέρον όλα τα σχόλια. Θα ήθελα εν συντομία να σας παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία ε, του σχεδίου έγκρισης. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επιμείνω ε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ακολουθήσει τα διαδικαστικά βήματα βάσει της νομοθεσίας και ότι και η ΕΦΣΑ έχει κάνει μια διεξοδική ανάλυση ε, κινδύνου σε ό,τι αφορά με τις ε, πιθανές παρενέργειες ή επιπτώσεις για την ε, ανθρώπινη και ζωική υγεία και το περιβάλλον. Βεβαίως ε, υπήρχε και η δυνατότητα υποβολής ε, παρατηρήσεων. Η ΕΦΣΑ απάντησε στα σχόλια και στις παρατηρήσεις και αιτιολόγησε την στάση της στην Διαρκή Επιτροπή. Βάσει και του κανονισμού 1829 σχετικά ακριβώ με αυτό το ζήτημα. Υπήρχε και δημόσια διαβούλευση για την γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ. Έχει αξιολογήσει τις ε, παρατηρήσεις η ΕΦΣΑ και δεν υπήρξαν νέα στοιχεία που να ακυρώνουν τη θετική γνώμη για αυτό το προϊόν. Βάσει των παραπάνω λοιπόν η Επιτροπή πρότεινε την έγκριση αυτών των ε, γάμματα και επισημαίνω και πάλι ότι αυτό συνάδει με τον σκοπό του κανονισμού για την διατήρηση και διασφάλιση ε, της Ζωή και υγεία ανθρώπων, ζώων και του περιβάλλοντο, αλλά και για, σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα του καταναλωτή. Η απόφαση ψηφίστηκε στα τέλη Ιανουαρίου και όπως ξέρετε δεν υπήρχε γνώμη περικατά και τώρα ε, υποχρεούται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει. Σε ό,τι αφορά τα επιστημονικά στοιχεία, η ΕΦΣΑ χρησιμοποίησε ένα πολύ συγκεκριμένο ε, γνώμονα ε, και συμπέρανε ότι και τα 20 αυτά, οι 20 υποσυνδυασμοί δεν ε, δημιουργούν κινδύνους και βασίστηκαν σε συγκεκριμένα δεδομένα αλλά και στοιχεία για επί πέντε υποσυνδυασμών. Έτσι απαντώ ε, σε αυτά που αναφέρονται ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία. Όχι, υπήρξε μία προσέγγιση με βάση τα δεδομένα από την ΕΦΣΑ. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια για τα ζενιοκτώνα, Πρέπει να θυμόμαστε ότι η έγκριση των ζυζανιοκτώνων ρυθμίζεται από, και διέπεται από την συγκεκριμένη νομοθεσία για τα ζυζανιοκτώνα και βέβαια ανάλογα με το κατά πόσο εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται ε, ένα εν λόγω το προϊόν που ετίθεται σε εμπορία θα πρέπει να τηρεί τα ε, μέγιστα όρια καταλήπων έστω ότι εγκριθεί ας πούμε ένα ζυνοκτόνο. το τελικό προϊόν θα πρέπει να σέβεται τα ε, ανώτατα επίπεδα καταλήπων που επιτρέπονται για αυτό το ζωνιοκτόνο. Εδώ, σε αυτό τον αραβόστο, δεν καλλιεργείται στην Ευρώπη, εισάγεται ω τροφή και ζωοτροφή. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι GMAs θα πρέπει να σέβονται τα ανώτερα επίπεδα καταλήπων που έχουν τεθεί για τα εν λόγω ζωνιοκτόνα. Εάν αυτά τα ανώτατα όρια τροποποιηθούν στο μέλλον, βεβαίω και αυτοί οι GMAs θα πρέπει να τηρούν και τα νέα επίπεδα όταν εισάγονται. Είναι σημαντικό λοιπόν να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ τη νομοθεσία γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών και ζενιοκτώνων. Ακόμα και αν στην πράξη οι GMAs αυτοί θα πρέπει να σέβονται τα ανώτερα, ανώτερα επίπεδα καταλήπων. Ακούσαμε βέβαια με μεγάλη προσοχή όλα τα σχόλια που ακούστηκαν σήμερα, όμως πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ακολουθήσει όλα τα βήματα της διαδικασίας και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να δεχθούμε ότι κατά οποιονδήποτε τρόπο έχουμε καταχαραστεί των εξουσιών μας, γιατί δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Ακολουθήσαμε όλη τη διαδικασία που προβλέπετε. Η ΕΦΣΑ έχει εκπονήσει ε, μια διεξοδικότατη ε, νομοδότηση. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να κατανοείτε γιατί ε, θεωρούμε αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη επιστημονικά ε, αυτή την ε, γνωμοδότηση και γιατί πιστεύουμε ότι και τα επόμενα βήματα είναι απολύτως νόμιμα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά θα ψηφίσουμε αύριο και στην Ολομέλεια στην 1 Απριλίου. Μάλλον στην 1η Ολομέλεια του Απριλίου. Ας προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο σημείο coming. It must be something <laughs> interesting. Um, another objection. Και άλλη ένσταση έχουμε τώρα. Αυτή τη φορά για το Triton 6%. Η κυρία Γκέρλινγκ έχει το λόγο ως εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η ένσταση διαφέρει από την προηγούμενη, ο λεγοντή, γιατί βασίζεται στο δικαίωμα ένστασης και όχι μόνο σε μια επιθυμία να πούμε κάτι. Πρόκειται για μια κατεξουδότηση πράξη που εμείς ως Επιτροπή έχουμε το καθήκον να εξετάσουμε και το δικαίωμα να ασκήσουμε ένσταση. Εγώ το έκανα γιατί με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα ε, ε, ε, ευρύτερα ο κλάδος ε, της φαρμακοβιομηχανίας υπήρχε μια γενικότερη ιδέα ότι όλες οι ουσίες ε, αυτές είναι κακές και τοξικές ουσίες. Όμως στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν πρόκειται για εγγενείς ιδιότητες αυτών των ουσιών, είναι πώς τις αξιοποιούμε. Και όταν αξιοποιούνται στον τομέα των, ε, επιστήμης έχουν σημαντικά ωφέλη για την ανθρώπινη υγεία. Ε, πρόκειται για ένα απολυματικό, ένα καθοριστικό για τα ε, φάρμακα. Ε, και αυτό μας δίνει ασφάλεια στον ιατρικό κλάδο και έχει λάβει την αδειοδότηση και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Χρησιμοποιείται σε φάρμακα για τον διαβήτη, τον καρκίνο, σε εμβόλια, σε διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ούτω καθεξής. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό αυτό το πλαίσιο όταν ε, ε, εξετάσει κανείς την ένσταση. Δεν νομίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ότι θα συνεχίσει να ε, χρησιμοποιείται ασφαλώς αυτή η ουσία σε αυτόν τον κλάδο και δεν νομίζω ότι είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει τέτοιες εγγυήσεις καθώς δεν έχει κάνει καμία ανάλυση κινδύνου συγκεκριμένα για τον τομέα της ανθρώπινης υγείας και των επιστημών αυτών. Ε, το θέμα είναι η διάρκεια της αδειοδότησης. Ενώ δεν προβλέπεται μέγιστη ε, περίοδος αδειοδότησης, θεωρία όμως, ε, θεωρητικά μάλλον, μπορεί να υπάρξει και ευρύτερη, πιο μακροσκελής αδειοδότηση, όμως de facto σήμερα η άδεια δίνεται για 12 χρόνια. Μια άδεια 12 ετής δεν λαμβάνει υπόψη τον κύκλο ζωής αυτών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπου μόνο οι κλινικές δοκιμές μπορεί να πάρουν 15 χρόνια. Οι επιχειρήσεις έτσι παίρνουν μια διοδότηση που δεν καλύπτει τον ε, πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων τους. Και αυτό γύρει ερωτήματα για τη βιωσιμότητα ε, του ευρωπαϊκού κλάδου και της παρασκευής αυτών των πολύτιμων προϊόντων. Επίσης, εφιστώ την προσοχή των μελών σε μια σειρά ασυνεπιών στην προσέγγιση της Κομισιόν. Όπως και στο εκτιμώντας F του ψηφίσματός μας, ε, εξαιρούνται από την οδοδότηση ουσίες που χρησιμοποιούνται στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αλλά όχι στην παρασκευή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Έτσι, η παρουσία, τα, ίχνη δηλαδή στο τελικό προϊόν εξαιρούνται, αλλά όταν χρησιμοποιείται η ουσία στην Παρασκευή δεν εξαιρείται. Ε, μου φαίνεται παράλογο και θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη της Κομισιόν εδώ. Έχω και άλλες όμως παρατηρήσεις. Δεν έχει αναπτύξει προσέγγιση η Κομισιόν σε σχέση με την ρήπανση από τα τεχνολογικά προϊόντα. Αν και γίνει αυτό, ίσως δεν θα χρειάζεται να κάνουμε τη σημερινή συζήτηση. Η Επιτροπή επίσης αδειοδοτεί ξεχωριστά την χρήση του Τράιτον ε, στην Παρασκευή υπό την αγροτική νομοθεσία. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι δημιουργεί οποιοδήποτε περιβαλλοντική ζημία η χρήση ε, της ουσίας αυτής. Και συγκεκριμένα προϊόντα που χρησιμοποιούν το Τράιτον δεν θα ε, πληγούν. Μόνο η ευρωπαϊκή βιομηχανία δηλαδή θα πληγεί ευρύτερα θα χρησιμοποιείται. Κλείνοντα, θεωρώ ότι η προσέγγιση τη Επιτροπή δεν ε, διασκεδάζει αυτέ τι σημαντικέ ανησυχίε, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι δυσανάλογη και δεν ε, ε, καλύπτει ε, του στόχου μα. Εκτιμώ ότι θέλουμε να προσθέσουμε ακόμα 11 ακόμα στοιχεία στο παράρτημα 14 όμως ε, θεωρώ ότι ήταν η επιλογή της Επιτροπής να ε, ομοδοποιήσει έτσι αυτές τις ουσίες και αυτό δεν μας έχει παρεμποδίσει στο παρελθόν. Και για την καφεΐνη είχαμε κάνει την ένσταση, όπου υπήρχε ακριβώς ο ίδιος αντίκτυπος ομαδοποίησης. Ε, περιμένω να ακούσω και τις απόψεις ε, των μελών και τις απαντήσεις της Επιτροπής. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στα μέλη. Σκιώδηση ή εκπροσωπή τους. Η κυρία Γκοστέτ πρώτη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να αντικαθιστώ το συνάδελφο Μαλού που απουσιάζει. Για να αποδείξω στους συναδέλφους ότι δεν είμαι καθόλου κατά των αντιρρήσεων αυτών, να τους πω ότι αυτή τη φορά θεωρώ ότι είναι τεκμηριωμένη η αντίρρηση αυτή. Επειδή Πιστεύω ότι αν στο παράδειγμα 14 του κανονισμού ΡΙΖ, δηλαδή τις πρώτες αδειοδοτημένες ουσίες, ουσίες οι οποίες να κάνουμε αυτό το τρίτον X100, θα ήταν λάθος. Με βάρος δημοσία υγείας, όπως είπε και η εισηγήτρια κυρία Γκέρλι. Χρησιμοποιείται λοιπόν σε δικασίες ε, κατασκευής διαφόρων ιατρικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων, ώστε να γίνει μια η απενεργοποίηση. Αν λοιπόν βάλουμε αυτό το τρίτο 100 χ στον κατάλογο των αδειοδοτήσεων ρις θα έχει επιπτώσει αυτό όσον αφορά άλλες βιομηχανικές διαδικασίες παραγωγής όπως οι βαφές. Και θα ήταν ε, πολύ κρίμα βέβαια και πολύ κακό αυτό για τη βιοτεχνολογία Βέβαια αυτή η απόφαση δεν οδηγεί στην πλήρη απαγόρευση αυτής της ουσίας. Θα υποβληθεί η χρήση της ουσίας αυτή σε μια προ-αδειοδότηση η οποία θα είναι περιορισμένη χρονικά, κάτι το οποίο όμως ε, ε, απειλεί να κάνει πιο περίπλοκες διαδικασίες και να μην επιτρέψει στις βιοεπιστήμίε ε, να έχουν νομική ασφάλεια, ασφάλεια δικαίου. Η διαδικασία λοιπόν αδειοδότησης αυτών των ουσιών συνήθως είναι μακροχρόνια και αν υπάρχει αβεβαιότητα, αυτή η αβεβαιότητα βεβαίως θα επηρεάζει την ανάπτυξη κατασκευασμάτων σε σχέση με το τρίτο εκατοχή. Και θα έχει βεβαίω επιπτώσει και στην παρασκευή συγκεκριμένων ιατρικών προϊόντων τα οποία δεν έχουν κανένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Βεβαίως να το λέξουμε αυτό, αλλά μην αφαιρεθούν, μην αποσυρθούν από την αγορά προϊόντα τα οποία δεν θέτουν κίνδυνο στην υγεία των ασθενών. Να εξετάσουμε λοιπόν τον κίνδυνο που παρουσιάζει αυτό το συστατικό. Συμφωνώ με την κυρία Γκέρλινγκ και αυτό θα έχει πει και ο συνάδελφο για τον οποίο μίλησα εδώ σήμερα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει πρόεδρο. Πορκ, έχει το λόγο. Ναι, ωραία. Συζητάμε εδώ επιτέλους τη σωστή αντίρρηση για αυτές τις ουσίες του παραρτήματος REACH. Στις βιοφαρμακευτικές ουσίες χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους η παρασκευή τους αυτή η ουσία αυτή τριτων και εκατό όπως είπαν οι προλαλήσασες. Πάντως η ΕΚΑ είπε ότι αυτή η ομάδα ουσιών έχει ενδοκρινολογικές επιπτώσεις όπως και οκταλφενόλες είναι επικίνδυνα χημικά αυτά με βλαβερές και σοβαρές παρενέργειες οπότε θα πρέπει να τεθούν σε αυτό το κατάλογο τώρα η χρήση αυτού του τρίτον χ100 βεβαίως έχει σημαντικές επιπτώσεις και στο περιβάλλον και το λέει αυτό και η Κομισιόν Οπότε δεν θα πρέπει να διατίθεται ελεύθερα στην αγορά αυτό το τρίτο και και θα πρέπει να υπόκειται σε διαδικασία διεδότηση. Η Κομισιόν λοιπόν προτείνει 20 ουσίες για το REACH, ουσίες οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται ευρέως και υπόκειται και αυτές σε αδειοδότηση. Αυτή, αυτός ο κατάλογος δεν σημαίνει βεβαίως όπως ακούσαμε προηγουμένως απαγόρευση αλλά απαγόρευση σε περίπτωση μόνο που δεν δοθεί άδεια. Αυτές λοιπόν οι ουσίες είναι επικίνδυνες σε σχέση με τις άλλες ουσίες τις οποίες, ε, τις οποίες έδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, Χημικών Ουσιών στις 6 του Φλεβάρου 14. Δεν χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε αδειοδοτήσεις οι οποίες θα είναι προβληματικές σε σχέση με το κατάλογο του παραρτήματος του ΡΙΤΣ. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, I have Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ριβαζή, βλέπω έχει ζητήσει το λόγο. Υπάρχει άλλος που θέλει να τοποθετηθεί γι' αυτό. Εάν όχι, κλείνω το κατάλογο των ομιλητών και δίνω το λόγο στην κυρία Ριβαζή. Τώρα. Πρώτα ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Γιατί πραγματικά πρέπει να κοιτάξουμε το πρόβλημα στα μάτια η Κομισιόν και τη συγχαίρω θέλει 12 ουσίες στο παράδειγμα 14 του Ρίτς λέγοντας ότι είναι ουσίες πολύ ενσυχητικέ που θα έπρεπε μελλοντικά να απαγορευτούν στην ε, ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ των τα θάλατα. Αν λοιπόν γίνει αποδεκτό αυτό, έχουμε 12 ουσίες οι οποίες θα απαγορευτούν και σε σχέση με αυτές τις ουσίες να πούμε ότι υπάρχει η LDT, e μια ουσία η οποία και αυτή παράγει το τρίτον χ100. Δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα. Είναι η υποβάθμιση αυτού του παράγοντα, του εντυγικού, που υποβαθμίζει σε οκτανιφενόλη και αποτελεί μία από αυτές τις 12 ουσίες που λέγαμε προηγουμένως και τις οποίες αφορά η απόφαση της Κομισιόν. Αν λοιπόν αποδεχτούμε την αντίρρηση της κυρίας Γκέρλινγκ, αυτές οι 12 ουσίες, οι οποίες είναι πολύ ενσυγητικές, δεν θα απαγορευτούν. Μου λέτε λοιπόν τότε ότι αυτός ο διοικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός για την ε, παρασκευή των πάντων ε, φαρμάκων, εντάξει, να το δεχτώ. Αν όμως αυτό ισχύει, τότε αυτό το LED, αυτό το εργαστήριο μπορεί να διαθέτει στην αγορά το τρίτον και η εταιρεία αυτή θα έχει στη διάθεσή τη 24 μήνες με φάκελο για να ζητήσει ακριβώς την παράταση της κρίσης. Οπότε το εργαστήριο θα μπορεί να το διαχειριστεί αυτό. Και το, το εργαστήριο θα πρέπει να θέσει τέλο πάντων ε, βέτο στη χρήση αυτών των ουσιών, στην απαγόρευση τη χρήση αυτών των ουσιών, ακριβώ για να προφλέξει τα συμφέροντά του. Αυτό όμω είναι απαράδεκτο. Αν ε, υπάρχει ένα εργαστήριο που θέλει να αναπτύξει ένα αντιοικό και έχουμε σημαντική υποβάθμιση, τότε θα πρέπει να ζητά αυτό το εργαστήριο συμπληρωματική αδειοδότηση. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα προϊόν το οποίο τέλο πάντων με τον τρόπο και τη διαδικασία που ακολουθούμε επιτρέπει τη χρήση των 12 ουσιών, οι οποίε θέτουν σοβαρού κινδύνου και ανησυχίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Λεκή Πρόεδρο. Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Απαντώντας στα επιχειρήματα της κυρίας Γκέρλινγκ στο σχέδιο του κειμένου, καταρχάς να πω σύντομα ότι δεν μιλάμε για κάτι εξουσιαδότηση εξουσιοδότηση πράξη αλλά κανονισμό που θα ακολουθήσει μια δικασία η οποία βέβαια ακόμα έχει προσαρμοστεί στα πλαίσια συνθήκη τη Λισαβόνα. Αντίθετα με αυτό που λέει η κυρία Κέρλινγκ, νομίζω ότι η αντιδότηση αποτελεί ένα προαπαιτούμενο στην πρώτη φάση χρήση αυτών των ουσιών. Και έχει σχέση με την, με την στο παράδειγμα του 14, του ΡΙΣ. Δηλαδή, όταν εντοπίζουμε μια ουσία που προκαλεί σοβαρέ ανησυχίε, τότε η διδιότησή του θα πρέπει να βασίζεται στι εγγενεί του ιδιότητε και λαμβάνοντα υπόψη τέλο πάντων του κινδύνου οι οποίοι προκαλούνται και η Κομισιόν αντίστοιχα θα πρέπει να αποφασίσει αν επιτρέπει ή όχι την χρήση. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αν μπορεί κανεί να λέξει του κινδύνου ή τέλο πάντων τα ωφέλη ξεπερνούν τα, τα πλεονεκτήματα, είναι περισσότερα τα μειονεκτήματα. Τώρα να σα πω, Πρόεδρε, την απόψή μα για τις ουσίες οι οποίες είναι εκτός αδειοδότηση δίσκη και είναι παρούσες σε ιατρικά προϊόντα και έχουν να κάνουν με το τρίτο και εκατό. Το ΡΙΤΣ υιοθετήθηκε με εξαιρέσεις για προϊόντα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια τη ε, διαδικασία παρασκευή. Και υπάρχουν άλλε ουσίε του παρακτήματο 14 που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση διαλυτικά ας πούμε, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή διαφόρων ιατρικών προϊόντων και που δεν βρίσκονται και αυτά στην τελική μορφή του προϊόντος και αυτά υπόκειται σε αδειοδότηση. Και υπάρχουν διάφορε άλλε αδειοδοτήσει οι οποίε διδόνται από την Κομισιόν για αυτέ τι ουσίε. Ή το ΕΚΑΣ, ας πούμε, ΕΚΑΣ έχει δώσει θετική γνωμοδότηση για τη χρήση του. Βεβαίω οι φαρμακοβιομηχανίε μπορούν να διαχειριστούν τη δικασία παρασκευής ε, μέσω του αιτήματος αδειοδότησης. Να πω επίσης ότι συμφωνούμε για τα 12 που ανέφερε η κυρία Αγγέλη προηγουμένως, 12 έτη. Το ΣΕΑΚ ως σύσταση στην Κομισιόν είπε κάτι αντίστοιχο, αλλά δεν υπάρχει στο κείμενο παρόμοια περιορισμό. περιορισμός. Μπορούν να δοθούν, ας πούμε, χρονικές περίοδοι πάνω των 12 ετών και επαφείται στις, αρχέ ε, αρχές των χωρών μελών όταν υπάρχουν λόγοι ε, για αδειοδότηση μεγαλύτερων χρονικών περιοδών από τις 12 ετίε, να δίδεται μια άδεια όπως έγινε σε μια περίπτωση όπου θεωρήθηκε κατάλληλο. Θα ήθελα επίσης να διορθώσω μια άποψη που ακούστηκε ότι οι άδειε υπόκεινται, δίδονται βέβαια για χρονικό, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά υπόκεινται σε επαναξιολογήσεις. Δεν έχουν λοιπόν απεριόριστη διάρκεια. Τώρα για την αβεβαιότητα και την έλλειψη προβλεψιμότητας που ανέφερε η κυρία Γκρόστετ. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακούμε συνεχώ από όλε τι επιχειρήσει, από όλου του κλάδου για όλε τι ουσίε που υπόκειται σε δικασία Και αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο εντάξει είναι αλήθεια, αλλά η Κομισιόν έχει καταβάλει σοβαρέ προσπάθειε για την ενίσχυση τη προβλεψιμότητα, ξεκινώντα καταρχά μια δημόσια διαβούλευση όσον αφορά την διάθεση στο εμπόριο και χρήση ουσιών πολλά χρόνια πριν την έναρξη αυτή τη διαδικασία. Κομισιόν λοιπόν κατέβαλε σοβαρέ προσπάθειε μαζί με την ΕΚΑ ώστε να υπάρχουν εγγυήσει για τι διαδικασίε αυτέ αναθεώρηση και επαναξιολόγηση, ώστε αυτέ να ισχύουν και να εφαρμόζονται. Ε, Βεβαίω, βελτιώνοντα την προβλεψιμότητα των ουσιών αυτών. Την διαδικασία αυτή την έχουμε διαχειριστεί πολλές φορές. Η κυρία Γκέρλινγκ είπε επίση ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης κινδύνου, ιδιαίτερα για αυτόν τον κλάδο. Αυτό ισχύει, είναι αλήθεια. Όταν έγινε η ανάλυση κινδύνου, έγινε αυτό επειδή οι αρχές δεν είχαν συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο και δεν είχαν δηλώσει τις ουσίες αυτές ως ε, επικίνδυνες στο κατάλληλο βαθμό. Όμως η ΕΚΑ έδωσε προτεραιότητα σε αυτές τις ουσίες και Κομισιόν ακολούθησε μια δημόσια διαβούλευση κοινωνικο-οικονομικού αντικτύπου, ενημερώνοντας για την χρήση και εξετάζοντα βεβαίω όλα τα επιχειρήματα της βιομηχανία. και κατέληξε στο ότι λόγω των πολλών υπολείπων χρήσεων αυτών των αδειοδοτούμενων ουσιών δεν υπάρχει λόγο να μην κάνει το ίδιο και η φαρμακοβιομηχανία επειδή ακριβώς δεν υπάρχει νομική βάση. Έχει περιορισμένο πεδίο, περιορισμένε δυνατότητε το ΡΙΤΣ να δώσει άδειε για συγκεκριμένου τομεί και νομίζω ότι υπάρχουν και απαραίτητε προποθέσει. Οπότε, έστω και αν τηρηθούν αυτά που προβλέπει το ψήφισμα, δηλαδή η πάυση τη χρήση, η, η ανάλυση κινδύνου κτλ. Θεωρούμε ότι πάλι στα ίδια συμπεράσματα θα είχαμε καταλήξει με αυτά που έχουμε μπροστά μα σήμερα. Και ένα τελευταίο σχόλιο προς την κυρία Ριβαζή. Δεν χρησιμοποιεί μόνο μια επιχείρηση αυτή την ουσία για την παραγωγή ιατρικών προϊόντων είναι διάφορες. Και για τα διαλυτικά που αναφέρθηκε προηγουμένως θεωρούμε ότι μπορούμε και εδώ να πετύχουμε επιτυχώς άδειε και τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν σε σχέση με αυτή την ουσία για την απενεργοποίηση δηλαδή των ιών κτλ. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την απόφαση τη ε, παροχής της άδειας και για την περίοδο επαναξιολόγησης τη ουσία. ουσία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε τη συζήτηση για αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Θα ψηφίσουμε αύριο. Και 1η Απριλίου Ολομέλεια. Επόμενο σημείο. Επόμενο σημείο, Λουλουσιεφ. Εξετάζουμε λοιπόν το σχέδιο έκθεσης. Ο εισηγητής είναι εδώ, κύριος Λίνς, και μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω το σχέδιο έκθεση σήμερα για το LULUCF, τον τομέα δηλαδή της ε, δασοκομείας, στα πλαίσια λοιπόν της ε, εφαρμογής της ε, Κλιματικής Συμφωνίας των Παρισίων. Όπως γνωρίζετε, στο Παρίσι υπήρχαν φιλόδοξοι στόχοι Και το σημαντικό είναι ότι σήμερα αυτή οι στόχοι θα είναι εφαρμοστές σε ένα εύρος τομέων και σε ό,τι αφορά τον Λουλουσιεφ επίσης. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τη γεωργία και την δασοκομεία. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε τον πρωτοποριακό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία του περιβάλλοντος και όχι μόνο αυτόν, αλλά και την συνεχόμενη ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιβαλλοντικά ζητήματα. Στο σχέδιο λοιπόν έκθεσης προσπάθησα να δείξω το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της γεωργίας και της δασοκομείας διότι ο τομέας αυτός είναι στο επίκεντρο πολλών πολιτικών, ε, πολλών απαιτήσεων, τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών, σε ό,τι αφορά την ε, παραγωγή τροφίμων, διάφορων σχετικών προϊόντων, δασικών προϊόντων, την βιώσιμη ανάπτυξη και πώς όλα αυτά επιδρούν στο περιβάλλον, στη γεωργία, στη δασοκομεία. Υπάρχει επίσης το θέμα της, ε, του διοξιδίου του ε, άνθρακα, της απορρόφησης ε, του διοξιδίου του άνθρακα από τα δάση, τα οποία είναι και το πρώτο θύμα της κλιματικής αλλαγής, μην ξεχνάμε. Είναι τα δάση αυτά που αντιλαμβάνονται πρώτα τις οποιασδήποτε κλιματικές αλλαγές. 9% λοιπόν είναι η τιμή την οποία συζητάμε. Πρέπει να υπάρξουν πρόσθετα κίνητρα έτσι ώστε να αυξηθούν αυτές οι τιμές. Τώρα σε ό,τι αφορά την ευελιξία του Λουλουσιέφ ε, για τον επιμερισμό της ευθύνης είναι κάτι ε, που βρίσκουμε θετικό. Πιστώσεις επίσης είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις πιστώσεις. Οι πιστώσεις δεν δίνονται αυτόματα, πρέπει να τις κερδίζουμε, γι' αυτό λοιπόν ε, πιστεύω πως ε, πρέπει να δίνονται κίνητρα και ανταμοιβέ για την σωστή ε, χρήση αυτών των πιστώσεων. Επίσης, ο κανόνας του no debit πιστεύω πως είναι κάτι που πρέπει να χαιρετήσουμε. Είναι ένας κανόνας που θα εφαρμόσουμε και στην LULUCF, ε, πέρα από την ενεργειακή πολιτική. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά ισχύουν μέχρι το 2030. Επίσης, η βιώσιμη διαχείριση των δασών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται να, δοθούν, να γίνουν επενδύσεις στην δάσωση, διότι δεν είναι μόνο η απορρόφηση του διοξιδίου του άνθρακα το όφελος που δίνουν τα δάση, αλλά πολλά ε, ακόμα, όπως γνωρίζετε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να εκμεταλλευτούμε αυτό το, την ανεξάντλητη δυναμική των δασών. Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι τα δάση στην Ευρώπη ε, χαρακτηρίζονται από μεγάλη πολυμορφία. Έχει να κάνει με το διαφορετικό κλίμα, με ε, τη γεωγραφία της ε, κάθε, χώρα, κάθε χώρας. Γι' αυτό πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις για τροποποίηση, για αλλαγή, υπάρχουν, σε αυτές, υπάρχουν στην έκθεση για παράδειγμα, αυτές οι δασικές τιμές αναφοράς, υπάρχει ένα καινούργιο χρονοδιάγραμμα που προτείνω από το 2000 μέχρι το 2012 η Κομισιόν προτείνει μέχρι το 2019 τη λήξη της ε, πρώτης ε, περίοδου. Ας μην ξεχνάμε πως το πρωτόκολλο του Κιώτο θα ισχύει μόνο μέχρι το 2019. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να πάμε πέρα από αυτό. και να φροντίσουμε οι στόχοι που θα τεθούν να είναι ε, εφαρμόσιμοι. Ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά αυτό το μοντέλο των τριών σταδίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να απλοποιήσει ε, τα πράγματα γυρίζοντας πίσω όμως Αυτές όμως, αυτά όμως τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων πρέπει να προσαρμόζονται ε, ανάλογα ε, το κράτος μέλος. Μετά, διαχείριση των δασών. Το όριο του 3,5% που προβλέπεται αυτή τη στιγμή για τις πιστώσεις προτείνουμε ιδιαίτερα για τα κράτη-μέλη που έχουν μεγάλες δασικές εκτάσεις, να γίνει πιο ευέλικτο. Να τους δώσουμε λοιπόν μεγαλύτερη ευελιξία. Γι' αυτό και σε αυτό το ποσοστό από το 3,5% στο 7% για ορισμένες χώρες όπως για παράδειγμα η Σουηδία ή η Φιλανδία που έχουν μεγάλες δασικές εκτάσεις έτσι ώστε να εγγυηθούμε μια ευελιξία. Μετά, είναι πολύ σημαντικό και το θέμα της δάσωσης και εδώ ε, οι πιστώσεις έχουν ένα ανώτατο όριο 20 ετών. Εμείς ε, προτείνουμε να μείνουμε σε αυτό το όριο και κατά εξαίρεση να υπάρχει μία ε, αύξηση στα 30 έτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως πιστεύω πως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γυρίσει προς τα πίσω στους στόχους της. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδες ηγητές και όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί μου και από άλλες επιτροπές, την ε, Γεωργία, την ε, Βιομηχανία, την Επιτροπή Ανάπτυξης, οι οποίοι συνέβαλαν πάρα πολύ στην κατάρτιση αυτού του σχεδίου έκθεσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λίντς. Το λόγο έχουν οι σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ. Τι χρόνο έχω στη διάθεσή μου για να μην τον υπερβώ. Έχετε χρόνο. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη σημασία ε, του κανονισμού Ρουλουσιεύ σε ό,τι αφορά το ευρύτερο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία εδώ για να συμβάλλουμε στην ευρύτερη διαδικασία της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που μας παρουσίασε ο Νόρμπερτ Λίνς ως εισηγητής θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική αφετηρία ε, υπήρξε πολύ συνεργάσιμος ε, στην όλη διαδικασία και νομίζω ότι η πρώτη φάση της επαφής ε, του εισηγητή με τους σκιώδεις ήταν ε, πολύ επικοδηματική. Πιο συγκεκριμένα τώρα από πλευρά Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να πετύχουμε με την ε, πρόταση αυτή για την χρήση γης, είναι τελικά να έχουμε καλής ποιότητας λογιστικά στοιχεία και θα επανέλθω σε αυτό, αυτό είναι το βασικό για μας. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το σημείο αναφοράς. Υπήρξε μια πρόταση από την Επιτροπή Περνόρμπριτ ότι προτείνεται ένα διαφορετικό χρονοδιάγραμμα ε, στη δική του πρόταση. Από πλευρά μα, εμεί θέλουμε να μην υπερβούμε το να μην πάμε πιο πίσω από το 2009. Γιατί μετά θα χαθούμε. Είναι σωστό αυτό που προτείνει η Επιτροπή. Αν πάμε πιο πίσω θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί το 2009 ε, υιοθετήθηκε η Οδηγία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αυτό άλλαξε τα πράγματα και νομίζω γι' αυτό ότι δεν είναι σωστό και γενικά οι σοσιαλδημοκράτες θεωρούν ότι δεν πρέπει να πάμε πιο πίσω από το 2009 το οποίο έχει επιλεγεί πολύ συγκεκριμένα ε, ως ε, τελικό σημείο. Δεν έγινε έτσι κατά τύχη. Ε, ετέθη το 2009 λοιπόν ως τελικό σημείο για τα λογιστικά στοιχεία γιατί τότε υιοθετήθηκε η οδηγία που προανέφερα. Μετά. Θέλουμε μέσα τη νομοθεσία αυτής να δώσουμε κίνητρα για την χρήση ξυλίας σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ξυλίας ε, μακροσκελούς ε, βίου, όπως αυτό εδώ το προϊόν που σας ε, παρουσιάζω εδώ, το οποίο θα αποτελέσει μια επανάσταση, θεωρούμε, στην Ευρώπη και στον κόσμο στα επόμενα δέκα χρόνια. Οι εταιρείε που παράγουν τέτοιου είδου υλικά, ιδίω στην Γερμανία, στην Αυστρία, έχουν δει αύξηση 25% πέρσι στις πωλήσει τους. Είναι ουσιαστικά το οικοδομικό υλικό του μέλλοντος. Και νομίζω ότι η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να δώσει κίνητρα ε, για την χρήση τέτοιου είδου ε, ξυλία στο μέλλον γιατί αποτελούν πολύ καλό υποκατάστατο για τον ε, χάλιβα και το τσιμέντο ε, που είναι πολύ ενεργοβόρα και καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες άνθρακα. Το ποσοστό τώρα σε ό,τι αφορά την χρήση γης και τους, τις καθαρές τιμές θα ε, μας απασχολήσει ιδιαίτερως. Η Επιτροπή προτείνει το 3,5%. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια καλή πρόταση, λογική. Ο κύριος Λίντς προτείνει να ανέβει στο 7%. Προτείνουμε εμείς χαμηλότερη τιμή, την τιμή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επανέρχομαι ε, στη σωστή λογοδοσία. Αυτό είναι ο βασικός μας στόχος. Το 3,5% ή το 7%, ό,τι και να είναι τέλο πάντων, δεν είναι το πώς θα επιβάλλουμε πολιτική ε, στις ε, επιμέρου ευρωπαϊκές χώρες. Να πούμε δηλαδή στη Φιλανδία ή στη Λετωνία, στην Αυστρία ή σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ποια πρέπει να είναι η πολιτική τη. Αυτό που λέμε είναι ότι χρειαζόμαστε ένα ομοιόμορφο ε, σύστημα το οποίο να ισχύει ε, λοιπόν για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για να μπορούμε να συγκρίνουμε και τα στοιχεία μας. Και εγώ νομίζω ότι η Φιλανδία, ας πούμε, δεν έχει ε, τίποτα που να τη φαίνει σε δύσκολη θέση. Αντιθέτως, ε, τα πηγαίνει και πολύ καλά. Και ναι, πράγματι σε ένα γράφημα βρέθηκαν στη μία άκρη του άξονα, γιατί δηλαδή απέχουν από τον μέσο όρο και καλό θα ήταν να το εξηγήσουν. Μπορεί να είναι επειδή το 80% της, ε, ε, της επικράτειάς της ε, αποτελείται από την εξηλία και γι' αυτό εντάξει, δεν μας προκαλεί έκπληξη ότι είναι πολύ αυξημένη η λοτόμηση ας πούμε σε αυτή τη χώρα σε σχέση με άλλες χώρες που θα έχουν λιγότερη ξυλία. Μπορούν λοιπόν πολύ εύκολα να εξηγήσουν τέτοιε χώρε όπω η Φιλανδία γιατί απέχουν από τι υπόλοιπε χώρε. Είναι θετικό λοιπόν παράδειγμα και δεν έχουν τίποτα κακό. Σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε που κατέθεσα για τον κανονισμό επιμερισμού των ε, βαρών, θα θέλαμε ω Σοσιαλδημοκράτε να υποβάλουμε κάτι και για τη Λουσιεύ. σε ό,τι αφορά την ε, υποχρεωτική χρηματοδότηση σε του υδροβιότοπους. Ε, αναγνωρίζουμε αυτόν τον τρόπο ότι ε, τα δάση ε, συμβάλλουν πάρα πολύ στην δέσμευση άνθρακα και θεωρούμε ότι οι υδροβιότοποι είναι ακόμα καλύτεροι ως προς αυτό. στην και στην Αγγλία ας πούμε, βλέπουμε ότι ε, συμβάλλουν πάρα πολύ στην απορρόφηση άνθρακα. Γι' αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα διαφυλάσσουμε αυτά τα μέρη και όπως και στο παρελθόν είδαμε και ότι έχουμε την ευκαιρία να ε, αποκαταστήσουμε ε, αυτά τα μέρη και γι' αυτό δεν θα πρέπει να ε, φυτεύουμε δέντρα στις, στους και θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι δεν θα γίνεται αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Άλλος και η εισηγητής τώρα. Η κυρία Βεσνεύσκα, δεν είναι εδώ όμως. Ο κύριος Σπίκα θα πάρει το λόγο εξ ονόματός της. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς, η κυρία Βυσνεύσκα ε, δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ σήμερα. Απέστειλε ορισμένα σχόλια, τα οποία θα σας επισημάνω σε ό,τι αφορά την έκθεση Λουλουσιέφ. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τον κύριο Λίντς για το σχέδιο έκθεσής του. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση παρότι υπάρχουν ακόμα ένα-δύο στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ενισχυθούν ή να προσδιοριστούν περαιτέρω. Ένα από τα πρώτα σχόλια αφορά τις ε, κατηγορίες ε, που απαρτίζουν ε, την νομοθετική πρόταση και πώς θα τα εξετάσουμε σε πλαίσιο εκτός ETS. Όλα αυτά βέβαια προσδιορίζονται στον κανονισμό, όμως θα πρέπει να τα εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Και βέβαια Έχουμε και τα επίπεδα αναφορά νοσοκομεία, ε, τα λογιστικά στοιχεία και τον έλεγχο των κρατών μελών. Όλα αυτά βέβαια θα πρέπει ε, να υπάγονται στην αρμοδιότητα του κράτου μέλου ε, και να μην παρεμβαίνει το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδίω ό,τι αφορά τον επιμερισμό των εξουσιών. αναφέρεται ένα ποσοστό και κατά πόσο αυτό θα πρέπει να αυξηθεί ή όχι. Αν μείνουμε ε, στο όριο που υπάρχει στην πρόταση, δεν νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει απαραίτητα σε ορθή διαχείριση των δασών. Και δεν ξέρω αν έτσι αυτό θα συνάδει και με το πνεύμα της Συμφωνίας των Παρισίων. Ελπίζω λοιπόν να λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις της κυρίας Βυσνεύσκα. Ο κύριος Τόρβαλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους Γερμινείς, γιατί θα μιλήσω γερμανικά σε αυτή τη φορά. Θα προσπαθήσω. Και όπως ε, μπορείτε να ακούσετε, ούτε τα αγγλικά ούτε τα γερμανικά είναι μητρική μου γλώσσα. Ε, καταρχάς θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας τον εισηγητή κύριο Λίντς. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με ένα πολύ τεχνικό θέμα και ε, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι διαφορετικά ε, κινδυνεύουμε να χάσουμε πάρα πολλά. Θα, θα χαθούμε στο δάσος κοιτάζοντας το δέντρο, για να παραφράσω την παροιμία. Αυτά λοιπόν ε, στα γερμανικά. Συνεχίζω στα αγγλικά και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πως το σχέδιο έκθεσης ε, δίνει έμφαση στην, ε, στις περιβαλλοντικές πρακτικές, χρησιμοποιεί τις εκπομπές διοξιδίου στα πλαίσια του Λουλουσιεφ. Όμως υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα. Το δάσος πόσο ακριβώς μπορεί να βοηθήσει στην απορρόφηση διοξιδίου του άνθρακα και υπό ποιες συνθήκες υπάρχουν κάποιες ελλείψεις ό,τι αφορά τα δικαιώματα εκπομπών ε, και πολλές φορές ε, ο κανονισμός Λουσιέφ χρησιμοποιείται ε, βοηθητικά, χρησιμοποιείται στην ουσία με τρόπο ώστε το δάσος καταλήγει να είναι το ζημιωμένο από όλο αυτό. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη ευελιξία στο σύστημα διότι πιστεύουμε πως αυτή τη στιγμή ε, δεν υπάρχει ισορροπία. Και από εκεί που κατάγομαι αυτό το αισθανόμαστε έντονα. Βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν προβλήματα και αν δεν προσαρμοστεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, χάσει οπαδούς. Αυτό το ανώτατο όριο λοιπόν του 3,5% που ε, αύξησε ο κύριος Λίνς, διπλασίασε στο 7% θα μπορούσε να ήταν ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Προσπαθήσαμε να δούμε πώς προέκυψε αυτό το 3,5%. Ζητήσαμε ε, πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από διάφορους οργανισμούς, όμως δεν πήραμε κάποια σαφή απάντηση. Και από ό,τι φαίνεται αυτό το 3,5% ε, το βγάλαμε από ένα καπέλο, το εμφανίσαμε από το πουθενά. Δεν νομίζω λοιπόν πως αυτός ο τρόπος είναι ο κατάλληλος για να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Η βιώσιμη δοσοκομεία είναι επένδυση για το μέλλον και η βιώσιμη γεωργία επίσης. Και πιστεύω ότι συμφωνούμε με τον εισηγητή, συμφωνούμε και με τους όλους συναδέλφους, ιδιαίτερα για την ε, υλοτόμηση, για, την ε, ε, για τα διαχειριζόμενα δάση και πιστεύουμε πως χρειάζεται να προχωρήσουμε και να εξελιχθούμε. Χρειάζεται λοιπόν να διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές ε, δασικής διαχείρισης σε άλλα ε, μέρη της Ευρώπης, όχι μόνο σε ε, λίγα. Γι' αυτό πιστεύω ότι και ο κύριος Λίντς και ο κύριος Μπρέναν έχουν παρόμοια άποψη με τη δική μου. Η σωστή δασική διαχείριση σίγουρα είναι κάτι θετικό. Επίσης, Πιστεύω πως καλώς τονίζεται ότι η δασική διαχείριση είναι ευρωπαϊκή υπόθεση και συμφωνούμε με τη σχετική παράγραφο στην έκθεση. Όμως έχουμε αρκετά προβλήματα με τα επίπεδα αναφοράς για τα δάση. Και αν δείτε το ιστορικό θα διαπιστώσετε ότι στη Φιλανδία ας πούμε άλλαξαν αυτά τα, ε, όταν άλλαξαν αυτά τα επίπεδα στα μέσα της δεκαετίας του 90 ας πούμε μειώθηκε ε, το τυράζ της εφημερίδες. Μετά υπήρχε το 2005 μια μεγάλη απεργία ένα μπλοκάρισμα και μια μεγάλη κρίση το 2009. Όλα αυτά επηρέασαν ε, τον τρόπο που υπολογίστηκαν αυτά τα επίπεδα αναφοράς και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί ένα δάσος και όλα αυτά που λέτε. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει ένα σαφέστερος ορισμός των πραγμάτων και να δούμε τι συμβαίνει στα δάση τα ίδια και όχι τι συμβαίνει στην κοινωνία. Όμως πιστεύω πως οι γενικές γραμμές ε, πάμε καλά. Προχωράμε σωστά, ιδιαίτερα μετά την ε, συνάρτηση των Τζίκωση στον Πάντεν Πάντεν. Νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ο μόνος μεγάλος ε, παράγοντας παγκοσμίω που θα αναλαμβάνει, θα έχει αναλάβει κάποιε ευθύνε. και αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Αν δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα σύστημα δασική διαχείριση. τότε δεν χρειάζεται να σα πω τι θα ακούσουμε από τον Τραμπ, τι θα πει. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω προ το παρόν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τόρβαλτς. Δεν κατάλαβα τι είπατε θα μιλήσετε γερμανικά, αυτό δεν το κατάλαβα. Μετά μιλήσατε αγγλικά, με μπερδέψατε. Κάποιο αστείο μπορεί να είπατε εσείς και να μην το κατάλαβα εγώ. Αλλά εντάξει, βλέπω πώ δεν βιαστήκατε. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριο Φλάναγκαν. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που άργησα γιατί έπρεπε να βρίσκομαι ταυτόχρονα και στην Επιτροπή Γεωργίας και μετά διαπίστωσα πως εδώ πέρα έχετε ε, δουλέψει πολύ γρήγορα. Ε, νομίζω πως ως ευρωβουλευτές προσπαθούμε να περάσουμε αυτές τις ιδέες τους αγρότες στην, Ιρλανδία, γενικότερα στην, ε, στους πολίτες και παρότι η πλειοψηφία μας συμφωνεί ότι σίγουρα πρέπει να γίνει κάτι για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα κτλ. Η κυριότερη ανησυχία μας είναι ο, στην Ιρλανδία ότι η τυρφώνες, οι, ε, τα έλλη, οι λόφοι, όλες αυτές οι περιοχές που για άλλους είναι άσχημες, για άλλους είναι ωραίες, θα πρέπει να δασωθούν έτσι ώστε να πιάσουμε αυτό το, αυτό το στόχο. Χρειάζεται λοιπόν, ε, πιστεύω, διαφορετική αντιμετώπιση στη λύση του προβλήματος. Αλλά αυτό υπάρχουν υπάρχουν και τα κατά. Τα κατά έχουν να κάνουν με αυτό που λέγαμε πριν. Εάν δηλαδή ένα δάσος είναι πραγματικά ε, μέρος που απορροφά ε, διοξίδιο του άνθρακα. Ε, να σας πω ότι στην Ιρλανδία πολλές φορές υπάρχουν δάση ατελείωτα και και στην Ευρώπη δάση ατελείωτα χωρίς ανθρώπους όμως πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Ε, αλλά τώρα, ε, σε ό,τι αφορά τους υγρότοπους και τους τυρφώνες, συμφωνώ να συμπεριληφθούν, αλλά είμαι λίγο επιφυλακτικός ως προς το, ε, τον εθελοντικό χαρακτήρα συμμετοχής κάποιων κρατών μελών. Ξέρετε, όταν γίνεται κάτι υποχρεωτικό, τότε οι πολιτικοί αρχίζουν και φωνάζουν ότι μας έδεσαν τα χέρια, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, αναγκαστήκαμε κτλ. Αλλά από την άλλη, όταν δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, όταν δεν είναι αναγκασμένος ένας πολιτικός να ε, αναλάβει ε, δράση, δεν κάνουν τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν μία μεσηλήση. Και ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι το εξή. Εγώ ε, είμαι από μια περιοχή πολύ πλούσια σε τύρφη. Το καλοκαίρι συλλέγουμε την τύρφη, πηγαίνουμε εκεί ε, και την τύρφη, ξέρετε, την κάνουμε καύσιμο. Υπάρχουν όμως κάποια προβλήματα Ε, και αυτά έχουν να κάνουν με αυτό που ακούω εδώ, ότι οι τηλεφώνε είναι άχρηστοι, δεν μπορούμε να του κάνουμε τίποτα. Ναι, μην ξεχνάτε όμω ότι υπάρχουν κάποιοι που ζεσταίνουν τα σπίτια του από αυτήν την τύρφη. Τι θα του πούμε τώρα, ε, φύγε από τη γη, δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, μπορεί να την κοιτά, έμενε αυτοί οι αιώνε, αλλά το σπίτι σου δεν θα το ζεστάνει από αυτή τη γη. Τι θα του πείτε, χρειάζεται αυτό, αυτές οι προτάσεις, αυτές οι ιδέες να συνδεθούν με ε, πρακτική σκέψη. Να δούμε ότι α, πολλές φορές αυτές οι προτάσεις μπορούν να ωφελήσουν τον ένα, αλλά θα διάσουν τις τσέπες του άλλου. Και θα αλλάξουν, όχι, και θα αλλάξουν επίσης και το, το περιβάλλον, την γεωγραφία της ε, χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάβορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα πρέπει να θεωρήσουμε τον κανονισμό Λουλουσιεφ μέρος ενός ευρύτερου ε, πακέτου, μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων που συνδεδεμένα με την ε, Σύμβαση των περισσίων στόχο έχουν να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Ε, αυτό λοιπόν είναι, αυτή η πρόταση που βλέπουμε εδώ είναι μόνο ένα μέρος της λύσης. Πρέπει να κοιτάξουμε με προσοχή τον κανονισμό Λουλουσιεφ και να δούμε αν πραγματικά συνεισφέρει στην επίτευξη αυτών των στόχων ή όχι. Επίσης, πρέπει να δούμε ποιους τομείς επηρεάζει ε, ο κανονισμός Λουσιέφ. Δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό το ζήτημα, είναι και θέμα βιοπικιλότητας, ε, είναι και θέμα άγριας ζωής, ε, δασικής διαχείρισης και γεωργικών δραστηριοτήτων, τυρφώνες που αναφέρθηκαν. Πρέπει να δούμε όλο λοιπόν ε, το θέμα, σε όλο του το εύρος. Τώρα η αρχική πρόταση της Επιτροπής από τον Ιούλιο του 2016 με τα ανώτατα όρια για ε, κάποιους κλάδους νομίζω πως δεν ήταν όσο φιλόδοξη έπρεπε ή μπορούσε να είναι υπάρχουν στόχοι, περιβαλλοντικοί, ε, πολύ σαφείς. Βλέπω βέβαια τα θετικά στοιχεία της έκθεσης του κυρίου Λίνς, ωστόσο πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης έτσι ώστε η έκθεση να είναι πιο αποτελεσματική προς την επίτευξη αυτών των στόχων. Ε, με λίγα λόγια πιστεύω πως την έκθεση πρέπει να προσθέσουμε και αυτήν την ευρύτερη εικόνα, να μην μείνουμε μέχρι το 2030, αλλά να ε, προχωρήσουμε πέρα από αυτό και να έχουμε κατά νου τους στόχους του 2050. Επίσης, άκουσα και ένα σχόλιο για τα επίπεδα αναφοράς με το 2009, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω πως αυτή η πρόταση είναι καλύτερη, διότι έτσι φαίνονται καλύτερα οι εξελίξεις στον ε, δασικό τομέα. Συμφωνώ λοιπόν με αυτή την πρόταση που, στην οποία αναφέρθηκαν για τα έτη 2000-2012. Τώρα είμαι εισηγητή στην Επιτροπή Ήτρε για έναν παρεμφερή κανονισμό και πράγματι βλέπω προβλήματα στην πρόταση για τον μηχανισμό ευελιξίας. Πιστεύω πως πρέπει να ξανακοιτάξουμε το θέμα για να βρούμε την ε, κατάλληλη συμβαστική λύση. Αναγνωρίζω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ε, αλλάξει, να επικαιροποιήσει τους κανόνες για τη λογοδοσία. Πιστεύω όμως ότι χρειάζεται διαφάνεια και ακρίβεια σε αυτόν τον υπολογισμό και πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε λοιπόν μια κατάλληλη μέθοδο. Μετά, η πρόταση πρέπει να συνεισφέρει στην σωστή χρήση της βιομάζας και να μην ξεχνάμε ότι η βιοενέργεια έχει άμεσες επιπτώσεις και στη βιοποικιλότητα. Θα υποβάλω βέβαια και γραπτά τα σχολεία και τις προτάσεις μου και θα ήθελα να ευχαριστήσω τέλος ξανά τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Εύη έχει το λόγο. Πρώτα ευχαριστώ. Να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή για τη δουλειά του. Όμως να σχολιάσω αντίστοιχα όπως έκανε και ο συνάδελφος προηγουμένως, ο κ. Γιάβορ. Παρόλο που λοιπόν αυτή η πρόταση εντάσσεται στο πακέτο μέτρων για τη μείωση κατά 40% των εκπομπών θερμοκηπίου στην Ευρώπη μέχρι το 2030, δεν θέτει στόχους αύξησης της απορρόφησης και περιορίζεται το συζύγιο των εκπομπών. Οπότε βλέπει εδώ ένας φιλόδοξος στόχος εκ μέρους της Κομισιόν στην πρόταση αυτή. Το LCF στην Ευρώπη πρέπει να συμβάλλει στην αφαίρεση 350 εκατομμυρίων τόνων ετησίως. Όμως οι, οι προβλέψεις μας μιλούν για μείωση, η υποχώρηση της απορρόφησης 2050 και μετά. Οπότε εδώ έχουμε να κάνουμε ακριβώς με, τις, με τη βιομάζα για χρήση παραγωγής ενέργειας. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να θεσπίσουμε δεσμευτικούς στόχους για το 30, το 40, το 50 με ξεκάθαρες στρατηγικές ενδείξεις για τους τομείς LLCF. και οι στόχοι θα πρέπει να ενισχυθούν. Άλλη μια πτυχή που μας ανησυχεί ιδιαίτερα αφορά την εφαρμογή στοιχείων ευελιξίας που ασχολούνται με τον Air Sharing. Η εφαρμογή αυτών των μορφών ευελιξίας θα πρέπει να οδηγήσει στη μείωση 38% των περικοπών προβλέπονται το 2050 σε σχέση με τον αρχικό στόχο του 40%. Οπότε εδώ διατρέχουμε το κινδύνο να μην πετύχουμε επουδενή τους στόχους που ήδη είχαμε θέσει. Θεωρούμε λοιπόν εμείς ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε οποιαδήποτε μορφή ευελιξίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κονδύλια που αφορούν τις περικοπές for sharing και να έχουμε ένα πιο αυστηρό κανόνα που να προβλέπει ότι η πώληση αυτών των πιστώσεων απορρόφησης θα επιτρέπεται για τις χώρες μέλη που δεν έχουν κάνει προσφυγή σε εργαλεία ευελιξίας όσον αφορά τους στόχους του for sharing. Διαφορικά νομίζω ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας κατάστασης αν όχι ατυχούς τουλάχιστον δύσκολες για τις χώρες μέλη. Και όπως είπα και άλλοι συνάδελφοι, θα πρέπει να έχουμε ένα νέο σύστημα για όλους τους τομείς που θα λαμβάνει υπόψη μόνο την ποσότητα σε έτος αναφοράς αποθηκευμένου διοξιδίου άθρακα. Και θα πρέπει επίσης να τονίσω ότι είναι απαραίτητο ο κανονισμός αυτός στο LULUCF θα πρέπει να αξιολογηθεί βάσει και των αντικτύπων στους στόχους για την διατήρηση της βιοποικιλότητας, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος η υποβάθμιση των στόχων διατήρησης της βιοποικιλότητας. Και τέλος, να πω ότι θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε τα κριτήρια βιωσιμότητας της βιομάσας για παραγωγή ενέργειας και να χρησιμοποιούνται μόνο για στόχους ή σκοπούς μείωσης των εκπομπών θερμοκηπίου. Αυτά που έλεγε προηγουμένω ο Σάφος πρέπει να βρίσκουν σύμφωνοι. Δηλαδή η μετάβαση προς ε, φυσικές ουσίες, ξυλία κτλ. και στον τομέα των κατασκευών, όσο πιο πολύ γίνεται αυτό, τόσο πιο πολύ θα έχουμε ωφέλη όσον αφορά την ε, εκπομπή διοξιδίου άνθρακα μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λέει πρόεδρος. Έχω ένα κατάλογο ομιλητών που θα κλείσω τώρα εκτός και αν υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει. Λίζα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τον Όρμπερτ Λίνς για τη δουλειά του και όσα έκανε στο σχέδιο έκθεσης. Πιστεύω πως είναι μια καλή βάση για εμάς εδώ στην Επιτροπή. Να αναφέρω τρία πράγματα μόνο. Καταρχάς, η δασοκομεία έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και όταν μιλάμε για προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα, όχι μόνο πώς θα επιτύχουμε τους ε, στόχους της ε, μείωσης κατά 1,5-2 βαθμούς της, της θερμοκρασίας του πλανήτη, αλλά και ε, να δούμε ότι η βιώσιμη δασοκομεία είναι καλή, καλή για το περιβάλλον. Χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην βιώσιμη δασοκομεία. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία ε, υπάρχουν μόνο στο χαρτί και δεν τηρούνται. Γνωρίζουμε όλοι ότι ε, τι έχει γίνει μάλλον με τα δάση και τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν, όπως αναφέρθηκε, διάφορες μέθοδοι υπολογισμού που ε, χρησιμοποιούνται, αλλά ε, αυτά τα έχουν ήδη πει άλλοι. Μετά, ε, δεν πρέπει να παραμελήσουμε ε, το σύνολο των περιβαλλοντικών δράσεων ε, δίνοντας έμβαση μόνο στα δάση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης σε κάποιες αντιφάσεις. Υπάρχει από τη μία διαπόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ETS. Εκεί δεν υπάρχει καμία ευελιξία. Υπάρχουν ε, ε, πράγματα που έχουν καταργηθεί, η καθαρή ανάπτυξη, οι κοινέ μέθοδοι αντιμετώπισης, όλα αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Από την άλλη υπάρχει, το, υπάρχει ο κίνδυνος της διαρροής άνθρακα και αν θέλουμε να τηρήσουμε αυτόν τον ε, φιλόδοξο στόχο του 43% δεν πρέπει να δείξουμε καμία ευελιξία. Τώρα στον επιμερισμό ε, των ευθυνών βρίσκω μόνο ένα 30% το οποίο δεν θεωρώ αρκετά υψηλό. Ε, νομίζω πως αυτό που θα γίνει είναι πως στο τέλος θα οδηγηθούμε σε ένα συμβιβασμό. Αλλά ας μην θυσιάσουμε την ευελιξία στο βωμό αυτού του συμβιβασμού. Αυτό δεν θα ήταν δίκαιο ούτε προς, τον, ε, προς ε, εκείνους που ασχολούνται και επηρεάζονται από το ETS, ούτε και για άλλους τομείς. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην υπερβούμε τα όρια που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να είμαστε δίκαιοι και στους άλλους κλάδους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ. Σύντομα. Γιατί υπόθηκαν πολλά. Πολύ σημαντικό το ζήτημα στα πλαίσια της εφαρμογής της Συμφωνίας των Παρισίων. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε περισσότερο τους κανόνες για τον υπολογισμό των εκπομπών και την αξιοποίηση των δασών για τη βιωσιμότητα και την ε, περιβαλλοντική ακριότητα του μηχανισμού. Υπολογίζουμε ότι χρειάζονται κάποιες διορθώσεις, αλλά η Κομισιόν πραγματικά για την χύση των δασών κάνει κάποιου υπολογισμού, δηλαδή βλέπει ας πούμε το τι κοπές είχαμε, τι ε, και η Κομισιόν για αυτά τα θέματα θα έχει την πλήρη αρμοδιότητα, κάτι το οποίο μου φαίνεται δυσανάλογο. Επιπλέον, για να καθορίσει κάποια επίπεδα, η Κομισιόν προτείνει να έχουμε ως αναφορά την περίοδο μέχρι το 2020, το οποίο σημαίνει ότι η δασοκομεία δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί, να είναι δηλαδή πιο έντονη σε σχέση με την περίοδο αυτή. Θεωρώ λοιπόν ότι για του εμπλεκόμενου στον τομέα τη δασοκομείας αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα και μια δυσκολία και θα επιθυμούσαν το επίπεδο αναφορά να είναι πιο εξελικτικό και να μην αφορά μόνο αυτή την περιορισμένη χρονική περίοδο. Και ο κόσμος της υπαίθρου και αγρότες εμπλέκονται. Δεν έχουμε να κάνουμε δηλαδή μόνο με τις μεταφορές ή τις κατασκευές και οι αγρότες καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες. Αν λοιπόν πρέπει να συμβάλλει και η γεωργία, δεν θα πρέπει να ζημιωθεί, γιατί πρώτος στόχος εδώ είναι η παραγωγή τροφίμων και όχι η παραγωγή τροφίμων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Είμαι βέβαιη ότι ο κύριος Λίντς, ο εισηγητής μας, τον οποίο στηρίζω με την έκθεσή του, με βέβαιος θα καταλήξει μια σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών των διαφόρων στοιχείων. Αυτά πρώτα ευχαριστώ. Και εγώ, κύριε Γκροστέτ. Σρέπρεκ, επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή κύριο Λίντ. μια πολύ καλή έκθεση. Τον ευχαριστώ για τι προσπάθειε του ε, για να καταλήξει σε αυτή την ισορροπημένη έκθεση. Εμεί ω κατοχώρε είμαστε υπέρ της διατήρησης κάποιης ε, σε αυτό το τομέα μεταξύ του κανονισμού ECR και αυτού, νου, ε, αυτού του κανονισμού, γιατί θεωρούμε ότι πρόκειται για μια θετική εξέλιξη και στον γεωργικό τομέα της δασοκομείας. Ε, βέβαια χωρίς να έρουμε και το κίνητρο ε, της καινοτομίας και σε άλλους ε, τομείς. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε θετικό κίνητρο στην διατήρηση των μηχανισμών μείωση των εκπομπών του άνθρακα. Βέβαια, πάντα με σεβασμό προς την βιοπικιλότητα. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία έρχεται πάντα αντιμέτωπη με, με μια μεγαλύτερη ζήτηση ε, για τροφή και τρόφιμα, Όμω, βέβαια πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου και την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγής. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά βέβαια, όμως θα πρέπει να παραμένουν και βιώσιμα και οικονομικά εφικτά. Και αυτό το ξεχνάμε εδώ κάποιες φορές. Το ίδιο ισχύει και για την νοσοκομεία. και στην χώρα μου και στην Γερμανία συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε ξυλία ε, για κάποιους ε, σκοπούς και θα πρέπει να το διατηρήσουμε και αυτό ως ε, μέσο αναφοράς. Πολύ συχνά μας έχουν απασχολήσει αυτά τα ζητήματα και πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Και τέλος, για τους ε, ε, κανόν, κοινούς κανόνες λογοδοσίας, θεωρούμε ότι συμβάλλουν στην επιτυχή εφαρμογή αυτών των μέτρων. Κυρία Γιούσου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο και του και ό,τι Να αναφερθώ μόνο σε λίγα στοιχεία. Καταρχάς, συζητάμε αυτή εδώ την πρόταση και αυτή για το for sharing ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα λοιπόν τα συζητάμε. Να ρωτήσω την Κομισιόν λοιπόν επειδή στην πρόταση για το force sharing υπάρχει μεγάλος αριθμός τροπολογιών. Προτείνουν 280 εκατομμύρια τόνων άνθρακα. για τις απορροφήσεις. Μου φαίνεται πολύ μετριοπαθής αυτός ο υπολογισμό. Πολλοί ζητούν περισσότερες, μεγαλύτερες ποσότητες, περισσότερους τόνους. Άλλοι ζητούν λιγότερους, τόνους βέβαια, αλλά νομίζω θα πρέπει να έχουμε περισσότερους τόνους. Οπότε να μου πει η Κομισιόν αν συμφωνεί με την αθεώρηση προς τα πάνω αυτού του στοιχείου ή αν θεωρεί αντίθετα ότι το μετροπαθέ επαρκεί για τις μορφές τώρα ευελιξία σε σχέση με τι απορροφήσει και τι αντισταθμίσεις. στι τωρινέ προτάσει επιτρέπουμε το υπόλοιπο της περίοδου 21-26 να πάει στην επόμενη περίοδο, 26 δηλαδή, 2030. Ρωτάω λοιπόν, αν οι εκπομπέ ή το υπόλοιπα εκπομπών αυτής της τελευταίας ε, περίοδου μπορούν να ληφθούν υπόψη για το 2030, ώστε να συνεχίσει να ισχύει το σύστημα. Μετά, για την ξυλία. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίε για να δούμε κατά πόσο αυτό το εργαλείο υπολογίζεται σωστά ή όχι οι εξισώσεις είναι περίπλοκες, οπότε θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό και να δούμε τι γίνεται ακριβώς με το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων ξυλίας και για την στάση μας για τις αγωγές εξαγωγές πρέπει να είμαστε αυστηροί. Τώρα, για τις φυσικές διαταραχές θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ο ορισμός των φυσικών διαταραχών επαρκεί και αν ο υπολογισμός του παρατήματος 6 είναι σωστός στατιστικά, ώστε να έχουμε ένα σωστό υπολογισμό αυτών των φαινομένων. Θα πρέπει ξαναλέω όμως να είμαστε αυστηροί και θα πρέπει να θεσπίσουμε κανόνες που θα είναι εύκολο να εφαρμοστούν για τους υπολογισμούς, αλλιώς θα καταλήξουμε σε καταστάσεις που θα προκαλέσουν γκρίνιες στη συνέχεια. Αυτά είχα εγώ να πω στα πλαίσια της πρότασης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η Πρόεδρος. Ο κύριος Ταντάν, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να χαιρετήσω καταρχάς τον συνάδελφο, τον συνάδελφο Λίσε για αυτή τη δουλειά που έκανε για το θέμα αυτό. Σε με τις περισσότερες θέσεις του, κυρίως για το επίπεδο αναφοράς και την επικουρικότητα. Ευελιξία επίσης, πιστώσεις, κονδύλια κτλ. Για το επίπεδο αναφοράς το εθνικό, όπως είπε σωστά και η κυρία Γκροστέτ, να εκφράσω και εγώ αμφιβολίες για το κατάλληλο επίπεδο από το 2009 και μετά. Νομίζω ότι οι υπολογισμοί ή τα στοιχεία αυτά θέλουν αμφιβόλω τη Συμφωνία των Παρισίων. Βλέπουμε ότι πρόσφατα έχουν εφαρμόσει οι χώρες μέλη μια βιώσιμη διαχείριση των δασών. Έστω και αν η Κομισιόν δεν έχει αρμοδιότητες για τα δάση. Νομίζω ότι οι χώρες μέλη είναι αρκετά ενεργές σε πολιτικές βιώσιμης διαχείρισης των δασών αφενός και αφετέρου. Νομίζω ότι σε σχέση με άλλες πολιτικές που έχουμε στην Ευρώπη και που εφαρμόζουν οι χώρες, όπως η βιομάζα για την παραγωγή ενεργείας, νομίζω ότι όλα αυτά έχουν ενταχθεί πολύ σωστά στις πολιτικές παραγωγής ενέργειας και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Αλλά από τη στιγμή που μιλάμε πολύ εδώ για κυκλική οικονομία θα πρέπει να προσέξουμε να είμαστε συνεπείς. Ένας συνάδελφος προηγουμένως μίλησε για τον άνθρακα και δεν μπορούμε να έχουμε πολιτική που αφενός ενθαρρύνει στις κατασκευές να έχουμε ολοκληρωμένα ξύλινα σπίτια αφενός και αφετέρου να έχουμε μια πολιτική που πλήττει τέλο πάντων εκμετέλευση των δασών. Πρέπει βεβαίω να διατηρηθεί το δάσο και η επιφάνεια, η δασική, σωστά εκμεταλλευμένη, να έχει κατάλληλη χρήση και κατάλληλο προορισμό για τρει, τέσσερι, πέντε γενιέ τέλο πάντων, αλλά με τα είδη που περιλαμβάνει το δάσο. Οπότε τα κριτήρια για τα επίπεδα αναφορά και τον ορισμό του δεν θα πρέπει να ακολουθούν αποκλειστικά και μόνο ιστορική βάση εξελικτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ταλτάν. Κύριε Τόρβολς, θέλετε να μιλήσετε. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα όμω, κύριε Τόρβαλτς. Γιατί έχετε ήδη πάρει το λόγο. Οπότε αν θέλετε μόνο εν συντομία ένα σχόλιο. Ναι, θα ήθελα μόνο να επισημάνω ότι έχουμε μελετήσει τον κανονισμό 525 κάθετος 2013 του 2013 που καθορίζει πώς θα πρέπει να υπολογίζονται τα επίπεδα αναφοράς. Και με αυτή τη βάση θα πρέπει να καταλήξουμε σε διαφορετική απάντηση από ότι αυτή στην οποία καταλήγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Βέλχαιμ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που κάνετε σήμερα. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ επικοδοματική και εξισορροπημένη συζήτηση αυτή που κάνουμε εδώ σήμερα. Να υπενθυμίσω ότι τα όσα πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι για την ε, πρόταση Λουσιεφ βασίζεται στα όσα έχουν ήδη συζητηθεί εδώ το 2012. Η πρώτη απόφαση Λουσιεφ συζητήθηκε λοιπόν τότε και Και αυτό πάλι μεταφράζεται όσα έχουν συμφωνηθεί ε, στο πρωτόκολλο του Κιώτο και έτσι μεταφέρονται στην ε, ε, ενωσιακή νομοθεσία. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της απόφασης αυτής και θα λέγαμε ότι τα κράτη-μέλη καταφέρνουν αρκετά καλά να υλοποιήσουν αυτούς τους λογιστικούς κανόνες. Το σημείο εστίασης βέβαια είναι ακριβώς αυτή, αυτά τα λογιστικά στοιχεία. Και έτσι είναι σημαντικό ότι η πρόταση Λουσιεύ και η πρόταση της Κομισιόν δεν προβλέπει νέε υποχρεώσεις για τους επιμέρους γεωργούς ή δασοκόμους και αυτό είναι ένα σημαντική πτυχή. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2014 ήταν μια σημαντική αφετηρία, γιατί αναγνωρίζουν και τις χαμηλότερες δυνατότητες ε, μετριασμού ε, για εκπομπές που δεν είναι ε, προέλευση, προέλευσης άνθρακα. Και με τον κανόνα No Debit, λοιπόν, με την ευρωπαϊκή πίστοση, αναγνωρίζουμε τις δύο όψεις νομίσματος, τις εκπομπές που δεν προέρχονται από τον άνθρακα αφενός, αλλά και αναγνωρίζουμε τη δυνατότητα κινήτρων για να συμπεριλάβουμε και την θετική όψη του νομίσματος, δηλαδή την βελτιωμένη ε, δέσμευση άνθρακα ε, και από άλλες δραστηριότητε. Επομένως, εξετάζουμε τα λογιστικά πρότυπα σε αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι σημαντικό για να διασφαλίσουμε ότι τα όσα περιλαμβάνονται ε, στα λογιστικά στοιχεία και στις πιστώσεις ε, των κρατών μελών είναι εύρωστα. Αυτό είναι σημαντικό. Οι λογιστικοί κανόνες ε, δεν ήρθαν από το πουθενά. Προέρχονται από το πρωτόκολλο του Κιώτο, το οποίο αποτέλεσε σημείο κίνησης για μας. θέλουμε βέβαια να τα επικαιροποιήσουμε, να τα απλουστεύσουμε, να τα ενισχύσουμε, για να έχουμε κοινά κριτήρια σε όλα τα κρατημέλη. Η πρόταση έχει ήδη αναπτυχθεί ε, στην Επιτροπή από κοινού και με το, από τον Επίτροπό μου, τον Επίτροπο Κανιέτε, αλλά και από τον Επίτροπο Χόγαν. και βλέπετε, το βλέπετε αυτό και από τον τρόπο που έχουν καθοριστεί οι μηχανισμοί ευελιξίας. Έχουμε βρει μια ισορροπία λοιπόν, τα 280 εκατομμύρια από τον ε, ένα κανονισμό στον άλλον συνδέονται με μια θεωρητική συμβολή ε, της ε, γεωργίας ε, non-CO2 και στην ε, καταπολέμηση των εκπομπών του άνθρακα και θεωρούμε ότι και η γεωργία αλλά και ο κλάδος Λουλουσιεφ παρέχουν κίνητρα και συμβάλλουν ε, στην ευρύτερη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, για κάτι συγκεκριμένα σημεία που αναφέρατε, η περίοδος ε, για αυτά τα επίπεδα, ε, το 3,5% που αναφέρεται και πάλι εδώ η αφετηρία μας ήταν αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή στην απόφαση Λουσιέφ και τα όσα εφαρμόζονται υπό το πρωτόκολλο του Κιώτο για αυτή την περίοδο. Όμως, βεβαίως είμαστε διατεθειμένοι να τα συζητήσουμε αυτά πιο εκτεταμένα. και ο ρόλος ε, των προϊόντων ξυλίας ε, στην οικοδομή θεωρούμε ότι είναι σημαντικός. Ε, μπορούμε να έχουμε πολλά υποκατάστατα και έτσι αναγνωρίζουμε και τα ωφέλη συγκεκριμένων προϊόντων ξυλίας. Θέλουμε βέβαια να δούμε πώς μπορούν να βελτιωθούν. Και Πιστεύουμε ότι τα ζητήματα βιοπικιλότητας είναι σημαντικά, δεν τα έχουμε αναφέρει σε αυτόν τον κανονισμό ερητός, γιατί έχουμε και άλλη κείμενη νομοθεσία στον τομέα της ε, βιοπικιλότητας, η οποία έχει πρέπει να γίνεται σεβαστή και γι' αυτό δεν την αναφέρουμε διεξοδικά. Χαιρετίζουμε και την χρονική συγκυρία αυτής της συζήτησης, γιατί προοδεύουν ε, οι συζητήσεις και στο Συμβούλιο. Επομένω, ε, θέλουμε να κινηθεί γρήγορα η διαδικασία και εδώ στο Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ την Επιτροπή. Ο εισηγητή, παρακαλώ, κύριε Λίντ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους στο σχέδιο έκθεσής μου. Νομίζω πως μπορούμε να δούμε πως αυτή η πρόταση για τον συγκεκριμένο τομέα της ε, δασοκομείας δηλαδή και της γεωργίας χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυμορφία και γι' αυτό είναι τόσο ε, περίπλοκη. Είναι κάτι διαφορετικό από το ETS και ε, αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε ή και να δούμε είναι πώς μπορούμε να μειώσουμε ε, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αλλά πώς θα γίνει αυτό δημιουργώντας ένα ευφυές σύστημα για μείωση των εκπομπών. Και όχι μόνο αυτό, πώς θα δώσουμε κίνητρα για ε, όσους ε, δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομείας να ε, εντείνουν τις ε, προσπάθειές τους προστασίας του περιβάλλοντος. Και συγκεκριμένα για την δασοκομεία υπάρχουν πολλά που πρέπει να δούμε ακόμα. Νομίζω πως και οι πολιτικές ομάδες μεταξύ τους θα χρειαστεί να συζητήσουν τα ανώτατα όρια, το 3,5% και αν θα προτείνουν κάποια αλλαγή. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά τα επίπεδα αναφοράς, νομίζω πως από αυτά που άκουσα υπάρχει μία σχετική συμφωνία. Αυτό τώρα που θέλω να πω είναι ότι με μεγάλη χαρά θα δω γραπτά αυτές τις προτάσεις σας, γιατί πιστεύω πως θα εμπλουτίσουν την έκθεσή μου. Θέλω να δω επίσης και τι θα πούν οι συνάδελφοι από τις άλλες ε, συνδεδεμένε επιτροπές. Γι' αυτό λοιπόν θα κλείσω εδώ και θα σας ευχαριστήσω ξανά. Ευχαριστώ και εγώ. 27 Μαρτίου είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τροπολογιών στις 11 το πρωί. Νομίζω πως εδώ ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας για σήμερα. Ναι. Δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα στην μερική διάταξη για σήμερα. Αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε. Προς το παρόν, καλό απόγευμα.